Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακαλώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, λοιπόν, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη, οι διερμηνείς μας με παρακάλεσαν να μας κάνουν μια σύντομη ανακοίνωση νομίζω ότι πρέπει να τους το επιτρέψουμε γιατί παίζουν έναν πολύτιμο και σημαντικό ρόλο. Έχετε το λόγο. Οι δερμηνείς σας πληροφορούν με τα λύπης ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις νέες συνθήκες εργασίας που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίησης για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα της διερμηνίας για τους ευρωβουλευτές και τους ευρωπαίους πολίτες κινδυνεύει. Δυστυχώ, λόγω της εργασιακής διαμάχης, η διερμηνία θα σταματήσει στις 12.30 ακριβώς, όπως προβλέπει το πρόγραμμα της συνεδρίασης. Ja, vielen herzlichen Dank. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ενημέρωση. Ελπίζουμε ιδιαίτερως ότι σύντομα θα υπάρξει μια σωστή ε, συμφωνία μεταξύ των διερμηνέων και της δίκης του Κοινοβουλίου. Όπως είπα, ε, μας παρέχεται μια απαραίτητη υπηρεσία και ξέρετε ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία σας και ότι χωρίς την συμμετοχή σας δεν θα μπορούσαμε να εργαστούμε. Οπότε να εκφράσω και πάλι τις ευχαριστίες μου, τις θερμές μου ευχαριστίες και σας εύχομαι επιτυχία στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις και συζητήσεις. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ημερήσια διάταξη. Λοιπόν, πρώτον, έγκριση τη ημερήσια διάταξη. Μπορούμε να κρίνουμε το σχέδιο ημερήσια διάταξη όπω έχει προταθεί. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Ωραία. Εγκρίθηκε. Λοιπόν, έχουμε έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Το σχέδιο ε, πρακτικών της συνεδρίασης της 25 Απριλίου είναι στα εγγραφά σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Ε? Οπότε θεωρώ ότι όπω συνήθω θα θεωρηθεί ότι ενεκρίθησαν τα πρακτικά αυτά εάν δεν υποβληθούν αντιρρήσει κατά τη διάρκεια της σημερινή μα συνεδρίαση. Λοιπόν, κατόπιν ε, ανακοινώσει ε, της Προέδρου. Σήμερα έχουμε διερμηνία για τις εξή ε, γλώσσε. Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Εστονικά, Ουγγρικά, Πολωνικά, Σλοβενικά, Βουλγαρικά και Ρουμανικά. Σα υπενθυμίζω, όπω πάντα, ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται ζωντανή στο ίντερνετ. Να περάσουμε τώρα στι αποφάσει των συντονιστών τη 16 η Μαου τρέχοντος. Οι αποφάσει των συντονιστών τη 16 η Μαου που εστάλησαν με email σε όλα τα μέλη της Επιτροπής θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί εάν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις μέχρι τις 22 Μαΐου. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι το προκαταρκτικό. Είμαι η Επιτροπή Πολιτισμού και Εκπαίδευσης και ε, προωθούμε ε, μια συγκεκριμένη άποψη αυτά. Ο Κούρτο Χόλσκι είπε στις 27 Ιανουαρίου 1919 ότι η σάτυρα πρέπει να υπερβάλλει και έχει δίκιο ε, τονίζει περισσότερο και υπερβάλλει την αλήθεια για να είναι ε, σαφέστερη. Τι είναι η σάτυρα λοιπόν, τα πάντα. Το θεωρώ ιδιαίτερα ε, απογοητευτικό ότι η πολωνική τηλεόραση 100 χρόνια μετά έχει άλλη άποψη και ε, έχει ε, υπάρξει δίωξη κατά της ε, σατυρίστριας ε, Κούρτς Κλάουντια Γιάχυρα με, γιατί ο λόγος ότι υπάρχουν ε, παραβιάσεις ε, πνευματικών δικαιωμάτων είναι φαινομενικός. Θα μπορούσαν να μπει και δύο μισή χρόνια φυλακή. πρέπει να ανησυχούμε όταν κάποιος λέει ότι και στον κομμουνισμό είναι δυνατό να περάσει κανείς στο δικαστήριο και να τιμωρηθεί. Θεωρώ ότι οι τελευταίες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα αρνητικές και πρέπει να επικριθούν δημοσίως. Ως Γερμανίδα και Ευρωπαία θεωρώ ότι είμαι υποχρεωμένη να το κάνω γιατί η Πολωνία ε, είναι πολύ σημαντική, είναι στην καρδιά όλων μας. Ήμουν εξίσου επικριτική για τις, ε, ε, τη συμπεριφορά των γερμανικών αρχών έναντι Γερμανών ε, σαντηρικών ε, που είχαν επικρίνει την τουρκική κυβέρνηση. Και θεωρώ ότι τα γεγονότα στην Πολωνία δεν έχουν διαφορετική φύση. Ελπίζω ότι μαζί με τους συναδέλφους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, Ραδιοφόρου και Τηλεόρασης θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους σατυρικούς καλλιτέχνες μας. Ε, αν δεν μπορούμε να γελάσουμε για τους πολιτικούς, τότε έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην ψηφοφορία και ψηφίζουμε για δύο ε, συγκεκριμένες γνωμοδοτήσεις. Ξεκινάμε με το σχέδιο γνωμοδότησης για την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών. Εισηγητής ο συνάλφος ε, Σαντιάγκο Φίσας. Δεν το βλέπω, άρα δεν μπορώ να το ρωτήσω αν θέλει να πάρει τον λόγο. Λοιπόν, έχουμε πολλές τροπολογίες ε, πήρα. Πήραν πολλές τροπολογίες επί των οποίων ε, διατυπώθηκαν 17 συμβιβαστικές. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τροπολογία 81. Α, όχι, δεν θα την ψηφίσουμε, είναι μόνο ε, γλωσσική. Οπότε περνάμε στο 82 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 86. Έχει αποσυρθεί. 87. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 88. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 103 έως 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Οπότε 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 108 έχει αποσυρθεί 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. Η 110 έχει αποσυρθεί. 114 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 115 και πάλι γλωσσική. Ωραία. 117 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 116 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 122 έχει αποσυρθεί και 124 ομοίωση συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 134 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 139 έχει αποσυρθεί η προφορική τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 18 συγγνώμη συγγνώμη ωραία να ελέγξουμε την 161 άρχεται Πέρας τη ψηφοφορια εγκρινεται Εγκρίνεται 13-10. Με συγχωρείτε, δεν ήταν σαφέ. Η 18 και 162. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. 163 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 164 για αποσυρθεί, 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 174 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9β υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 193 υπέρ. Κατά αποχές Α, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Είναι 103 ε, πίπτη, 192 λοιπόν υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 194 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 202 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές δεκτή 203 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 έχει αποσυρθεί 206 υπέρ κατά αποχές δεκτή 207 υπέρ κατά αποχές δεκτή 28 και 209 υπέρ κατά αποχές δεκτές 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά άποχες δεκτή 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή Λυπάμαι. Στην, πάμε στην προφορική τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Λοιπόν, σας παρακαλώ να επαναλάβουμε. 2.14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 2.15 υπέρ. Κατά αποχές Απορρίπεται. 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.16 και 2.17 ταυτόσιμες υπέρ κατά Λοιπόν, να τις ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. 14-11 εγκρίνεται. Εγκρίνονται. Οπότε πάμε 35. Ε, κάποιες σελίδες παρακάτω. 35. Τη βρήκατε. 35 λοιπόν υπέρ. Κατά. Α... Λοιπόν, επαναλαμβάνω. 35 στη σελίδα 17 τουλάχιστον στο δικό μου κατάλογο. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω το απορρίφθηκε, αλλά ελέγχουμε. Άρχεται. Πέρας. Ναι, 15-10 απορρίπτεται. 36 ε, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά Αποχές δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Όχι, συγγνώμη, 45, 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται για να έχει αποσυρθεί 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ελέγχουμε άρχεται την 47 ε. πέρας 11-14 Απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 14 έλεγχα. Λοιπόν, οπότε περνάμε στη συμβαστική 13. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται 21 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, μία αποχή, την πλειοψηφία. Συγχαίρουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Οπότε περνάμε στην ε, γνώμοδότηση για το σχέδιο προπολογισμού του 2019 και την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Ο συγκητή μα ήταν ο Μόρτεν Λόκεγκαρτ. Μόρτεν, θε να πει τίποτα. Απλώ για την τροπολογία 27 ότι αποσύρεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Λοιπόν, να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. απόχέ Δεκτή. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 7. Υπέρ. Για την 7 λέω. Υπέρ παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχέ, δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχέ, δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. απόχέ, δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. αποχέ. απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. απόχέ, δεκτή. 27 έχει αποσυρθεί λοιπόν. 28. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Ωραία. Δεύτερη παράγραφος τώρα. Τις 28 λέει πρώτος υπέρ. Πέρας. 14-9 εγκρίνεται. Λοιπόν, 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Προφορική 2 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 32 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 33 υπέρ. Κατά αποχέ, δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές να την ελέγξουμε την 36 άρχεται πέρας 11-12 απορρίπτεται. 37 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι ήταν ε, ο ίδιος συσχετισμός, αλλά ας το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 37 άρχεται. Πέρας. 9-12 απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ονομαστική άρχεται. Πέρας. 19 υπέρ, καμία ψήφος κατά και τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν ομόφωνα. Συγχαίρουμε τον εισηγητή και το ευχόμεθα κάθε επιτυχία στις περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Οπότε ολοκληρώνονται οι ψηφοφορίες και περνάμε απευθείας στο επόμενο θέμα που είναι το 6. Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης η κοινωνική και ε, πολιτική απασχόληση στο χώρο του ευρώ. Εισηγητής ο κύριος ε, Χουντής, ε, τρόπο μέχρι τις 12 Ιουνίου, 11 το πρωί και η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Ιουλίου. Λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Χουντή, 5 λεπτά για την παρουσίαση. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, ναι, περιμένω λιγάκι για την ησυχία της αίθουσα. Άλλωστε η αίθουσα είναι μεγάλη, μας έχει σε απόσταση και <laughs> δυσκολεύεται λίγο η επικοινωνία, ίσως και έτσι. Ευχαριστώ πολύ, εν πάση περιπτώσει, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι το θέμα της συγκεκριμένης γνωμοδότησης που μου αναθέσατε είναι σημαντικής εξέχουσα σημασίας για τη ζωή και την καθημερινότητα των κατοίκων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ η Επιτροπή μας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πώς επιδρούν η δομή και οι κανόνες της ΟΝΕ στις πολιτικές για την εκπαίδευση των κρατών μελών και κατά συνέπεια στις κοινωνικές πολιτικές της Ένωσης και τις πολιτικές απασχόλησης. Η εφαρμογή της ΟΝΕ στην πράξη είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και την επιπλέον διαίρεση μεταξύ πλούσιου βορρά και φτωχού νότου οι κανόνε τη Ευρωζώνης απαγορεύουν στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν το μείγμα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών που αυτά επιθυμούν σύμφωνα με τι ανάγκε των λαών του. Οι προπολογισμοί των κρατών μελών πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την Κομισιόν ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τι πολιτικέ κατευθύνσεις που αυτή έχει επιλέξει. Εν τέλει, η τήρηση των εξαντλητικών και κοινωνικά παράλογων, κατά την άποψή μου, κανόνων τη οικονομική διακυβέρνηση, και του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται με εμφατικό τρόπο τα τελευταία, την τελευταία δεκαετία, έχουν πλήξει σοβαρά τον τομέα της εκπαίδευσης και τις κοινωνικές πολιτικές στο σύνολό τους, τα κράτη-μέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πολιτικές λιτότητας που εφαρμόστηκαν στα περισσότερα κράτη της Ευρωζώνης έχοντας ως στόχο τη θωράκιση του ευρώ βασίστηκαν στη μείωση των δαπανών για την εκπαίδευση, την υγεία, τον πολιτισμό, της πολιτικές απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Ως αποτέλεσμα, με το μείγμα αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονταν στην Ευρωζώνη, στις στα περισσότερα κράτη-μέλη οι πολιτικές εκπαίδευση έχουν υποβαθμιστεί. Η δημόσια εκπαίδευση υποχρηματοδοτείται, το ποσοστό των κοινωνικά αποκλεισμένων πολιτών αυξάνεται, το ποσοστό, το φαινόμενο, του brain drain της ε, μετανάστευσης, δηλαδή εγκεφάλων, διωγγώνεται ιδιαίτερα από τι χώρε του Νότου. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν δομηθεί με κυρίαρχο σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών τη αγορά-εργασία και όχι την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη των συμμεταχόντων. Το κείμενο λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ζητά στο πλαίσιο λοιπόν της γνωμοδότησής μας την αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, υποστηρίζει την ίση πρόσβαση για όλους στην ποιοτική εκπαίδευση και σε ευκαιρίες διαβίου μάθηση, τονίζει την ανάγκη για μια γνήσια αναθεώρηση των πολιτικών για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τις δεξιότητες με επίκεντρο το συμμετέχοντα και όχι τις επιταγές των αγορών. Όλα τα παραπάνω, αγαπητοί συνάδελφοι, προσπάθησα να τα τοποθετήσω στον περιορισμένο χώρο που μου επιτρέπει ο κανονισμός. Ε, δεν θα σας παρουσιάσω κάτι παραπάνω αναλυτικό, είναι υπόψη σας. Ε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Γραμματεία της Επιτροπής μας για τη βοήθεια στη σύνταξη και στην ε, τεκμηρίωση της γνωμοδότησης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και περιμένω τις δικές σας παρατηρήσεις για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Χουντή για την παρουσίαση της γνωμοδότησής σας. Να περάσουμε τώρα στους σκιώδεις. Η Ζαμπίνε Φεχάιεν που εκπροσωπεί τον Σάλφο Ζαγοράκη. Ευχαριστώ. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του κυρίου Ζαγοράκη που δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ. Υπήρχαν άλλε συνεδριάσει τι οποίε έπρεπε να παρευρεθεί. Εκ μέρου του θέλω να πω ότι η βάση του κειμένου είναι καλή. Ο κ. Σκουντή έχει αναλύσει τι κοινωνικέ και οικονομικέ ανισότητε στην Ευρωζώνη με καλό τρόπο και έχει επισημάνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει την ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση, παιδεία και διαβίου κατάρτιση σε όλους. Ε, για μας το ΕΛΚ είναι σημαντική για την απασχολησιμότητα των Ευρωπαίων, ιδίω των νέων όλα αυτά. Ε, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε την απαραίτητη μέρημνα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που να συνεργαστούν αποτελεσματικά για να δημιουργήσουν καλύτερε ευκαιρίε μέσω τη εκπαίδευση και τη παιδεία. Και θα πρέπει να βοηθήσουμε με προγράμματα μαθητεία, άσκηση, παρακολούθηση και να συμμετάσχουν περισσότεροι δάσκαλοι, επιχειρηματίε, μαθητέ και φοιτητέ των προγραμμάτων Εράσμου. Βάσω του Ευρωβαρομέτρου κάθε, ε, μάλλον ένα στου δύο νέους από τα 18 έως τα 35 είχε μία τουλάχιστον εμπειρία ε, μαθητείας. Ένας από τους 10 πρώην μαθητευόμενους ξεκίνησαν τη μαθητεία τους μάλλον δήλωσαν ότι η περίοδο μαθητεία του ήταν ε, πολύ χρήσιμη για να βρουν μια κανονική θέση εργασία. Η μελέτη αυτή δείχνει ότι οι ποιοτικέ ε, ασκήσει και μαθητείε μπορούν να διασφαλίσουν πρόσβαση σε επαγγελματική αποκατάσταση. Γι' αυτό στηρίζουμε την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία όπω την εγγύηση για του νέου και την ε, πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να εγκρίνουμε αυτού του μηχανισμού και να γίνουν περισσότερο ε, προσβάσιμη σε όλους. Η ε, φυγή των ε, ταλαντούχων νέων ε, ιδίω στι νότιε χώρε, είναι ένα σημαντικό φαινόμενο. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματικέ στρατηγικέ για τι πολιτικέ εκπαίδευση και κατάρτιση, δίνοντα κίνητρα στου νέου για να επενδύσουν λόγω χάρη στι δυνατότητε επιχειρηματικότητά του. Ω ε, Επιτροπή Πολιτισμού, πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στην ε, αντιμετώπιση τη έλλειψη απασχόληση για όλου του εργαζομένου και να στηρίξουμε τον τομέα των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δημιουργών. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε μέρη για να διασφαλίσουμε εργασιακές συνθήκες για όλους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Ζαγοράκης ως και όδης του ΕΛΚ θα υποβάλει κάποιες σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πρόεδρε. Εξ ονόματο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσω με όσα είπε ο συνάδελφο Βεχάρεν και θα συγχαρώ τον εισηγητή με τον οποίο συμμεριζόμαστε τις ίδιες βασικές μέρημνες. Έχοντας υπόψη το, ότι το αντικείμενο της γνωμοδότησή μας είναι η ανάλυση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, όπου έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή Πολιτισμού, και επειδή μιλάμε για τις 19 χώρε της Ευρωζώνης, είναι σαφές ότι οι κατευθυντήρε γραμμές που θα πρέπει να κατευθύνουν τη συζήτησή μα, είναι αυτές που αναφέρονται και περιλαμβάνονται και στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Θεωρώ ότι δύο τα βασικά θέματα στα οποία πρέπει να σταθεί η Επιτροπή μα και να παρέμβουμε επί τη ουσία η εκπαίδευση από την παιδική ηλικία στο πανεπιστήμιο και η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην εργασία, στον επαγγελματικό χώρο. Είναι σαφέ ότι μια ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση πρέπει να ξεκινάει από το εκπαιδευτικό σύστημα και εκεί να έχουν πρόσβαση όλοι, ώστε να μπορεί ο καθένα να αναπτύξει τι δεξιότητε και ικανότητέ του, ανάλογα βεβαίω με το τι ταλέντα έχει και κλήσει ε, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ετησίω, όπω ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει μια κοινή ε, μελέτη για την εκπαίδευση, όπου αξιολογεί τι επιδόσει των κρατών μελών μέσω ενό ε, συνόλου δικτών, που από το 2018 θα είναι σημείο αναφορά και στο λεγόμενο ε, κοινωνικό βαθμολόγιο. Οι δείκτε αυτοί μετρούν λόγω χάρη των αριθμό των ανηλίκων που έχουν πρόσβαση στι υπηρεσίε για την επιακή ηλικία ή την παιδική ηλικία, τα αποτελέσματα των μαθητών στου διαγωνισμού τη ΠΙΖΑ, όπως και την πρόσβαση στην ε, το βάθμιο εκπαίδευση. Αυτοί οι δείκτες ε, θα πρέπει να είναι ώστε δυνατόν ακριβέστεροι και να συμπληρωθούν, διότι αποτελούν τη βάση για τις ειδικές συστάσεις ανά κράτος που κάθε χρόνο ε, δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να πω ότι προσφάτως διαπιστώθηκε από σχετικές μελέτες ότι υπάρχει σύνολο δικτών με κάποιους περιορισμούς. Το εντόπισαν η ΕΤΟΚ και η ΕΟΚΕ, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. Ε, γι' αυτό λοιπόν σε σχέση με το κείμενο που μας έστειλε ο ε, συνάδελφος Χουντής σκοπεύουμε να ε, υποβάλουμε κάποιες άμεσες αναφορές στο σύστημα δικτών που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ακριβώς με στόχο να γίνεται μια πιο ακριβής ε, και σκόπιμη καταμέτρηση. Ε, στις προτάσεις αυτές θέλω να προσθέσω και τα εξή. Ε, κάποια πιο συγκεκριμένα αιτήματα. Να υπάρξει κατάλληλη χρηματοδότηση στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 για την εγγύηση των νέων, ε, ανάλογα με τι αρμοδιότητέ μα βεβαίω. Ε, μια πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων που πρέπει να συνεχιστεί και εδώ να είμαστε λίγο πιο ε, συγκεκριμένοι και όχι πολύ γενικόλογοι. Δημόσιε και κρατικέ επενδύσει, εθνικέ επενδύσει για την εγγύηση των νέων και την συμπερίληψη των νέων στην αγορά εργασία και όλα αυτά σε έναν κανόνα για την κοινωνική συμμετοχή και στα πλαίσια των όσων επιτρέπει το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Εδώ η ιδέα είναι ότι αν θέλουμε μια σοβαρή παρέμβαση ε, στον κοινωνικό τομέα πρέπει από τη μια να αυξήσουμε τα κονδύλια που διαθέτουν τα εργαλεία αυτά και έπειτα να δείξουμε μεγαλύτερη ευελιξία στι δαπάνε των κρατών μελών ε, για να υπάρξουν κρατικέ δαπάνε από, μέσω δαπανών επενδύσεων μάλλον στο ανθρώπινο κεφάλαιο για να ολοκληρώσει κοινωνική πολιτική στην Ευρωζώνη πρέπει να περάσει και από συγκεκριμένε επενδύσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και με πολιτικέ για τη στήριξη τη παρακολούθηση των νέων από την παιδική ηλικία στο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι η Επιτροπή του Πολιτισμού θα καταφέρει να πετύχει μεγάλη συνέχεια συνένεση εδώ για να έχουμε μια ισχυρή έκθεση σκόπιμη με την όλη μας μελέτη του θέματος. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους του ECR και των φιλελευθέρων δεν έχουμε παρόντες τους σκιώδης ηγητές από το EFTD. Α, μόλις έφυγε από την αίθουσα ως και ο αντισηγητής της EFTD. Κυρία Μπίλντε, δεν ξέρω αν θέλει το λόγο. Θέλετε το λόγο, κυρία Μπίλντε. Εκτός μικροφώνου, δυστυχώς, τα σχόλια της κυρίας Μπίλντε. Okay, Σας ευχαριστώ. Να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε τσεχική καμπίνα γιατί κάποιος ασθένησε. Βέβαια, μπορείτε να μιλάτε τσεχικά, αλλά δεν μπορείτε να ακούτε την τσεχική διερμηνία. Ε, φαίνεται ότι και με την Ουγγρική διερμηνία υπάρχει πρόβλημα. Ούτε παθητικά, ούτε μπορεί κανείς να μιλά ε, Γκρικά. Ευχαριστούμε κυρία Κώστα. Ε, ευχαριστώ. Θα συμφωνήσουμε πολλά όπως είπε ο κύριος Μόργανο. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότεροι στην έκθεση αυτή, διότι βρισκόμαστε και στι παραμονέ τη εφαρμογή νέων πολιτικών στα πλαίσια του πολιτικού δημοσιονομικού πλασίου και μια από τις βασικές, ένα από τα νέα κοινά στοιχεία είναι τα καινούργια κριτήρια για τι πολιτικέ τη συνοχές που έχουν συμπεριληφθεί και στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματο, τη εκπαίδευση ε, ε, των πολιτών. Είναι σημαντικό λοιπόν να κάνουμε ένα πρώτο βήμα εδώ, αυτό που ανέφερε πριν και ο κύριο Μόργανο, κάτι που έχουμε ζητήσει πολλέ φορέ. Οι επενδύσει των κρατών μελών στο εκπαιδευτικό σύστημα, ιδίω στι ε, μειονεκτούσε περιοχέ, να ε, βγουν από το Σύμφωνο Σταθερότητα. Να θεωρούνται έστω επενδύσεις στην καινοτομία και την τεχνολογία. Ε, είναι λοιπόν σημαντικό εδώ να δούμε την υποχρέωση των κρατών μελών να εφαρμόζουν καλύτερε εκπαιδευτικέ πολιτικέ, ιδίω σε στιγμέ και περιόδου κρίση, αλλά και η διαβίου μάθηση να ευνοήσει τι πολιτικές παρακολούθησης και στήριξης με υποτροφίες ενδεχομένως, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχει λιγότερη ε, εγκατάλειψη του σχολείου και δεύτερες ευκαιρίες σε νέους, σε παιδιά που είναι ακόμα πάρα πολλά και βρίσκονται σε, δύσκολες, ε, σε δύσκολη περίοδο, αυτά να τα στηρίζουμε με τη διαβίου μάθηση. Επίσης, σωστά λέει ο εισηγητής, ότι πρέπει να υπάρχει περισσότερο εθελοντική συμμετοχή και όχι ε, αυτό που συμβαίνει τώρα, να υπάρξει αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων, των γλωσσικών δεξιοτήτων, των ε, μαθητιών και ασκήσεων, με την αγγίση των νέων και ίσως με μια ηλεκτρονική ε, κάρτα για τους ε, Ευρωπαίους νέους και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που να πολλαπλασιάσουν τις δυνατότητές τους να είναι κινητική στο εκπαιδευτικό σύστημα με τρόπο πιο συγκεκριμένο, πιο χειροπιαστό. Και να ολοκληρώσω ω προς τα Η εκπαίδευση σκοπό δεν έχει μόνο να βρει απασχόληση σε κάποιον, αλλά να επιτρέψει και την προσωπική ανάπτυξη για να έχουμε ε, πολίτε ελεύθερου και να μπορέσουν με τον καιρό, αν χρειαστεί, να αλλάξουν και δουλειά. Äh, Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε, ήταν παρανόηση. Ε, αν θέλετε, παρακαλώ έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εισηγητή. Η επένδυση στην ανώτατη εκπαίδευση πολλές φορές εξαρτάται από, ή μειώνεται από την φυγή των ε, ταλέντων, τις πολιτικές ελιτότητες και ε, μερικές φορές διευκολύνεται από τις διαδικασίες της Μπολόνια και του Εράσμους. Έχουμε μια εργασιακή μετανάστευση. Μια Ολλανδική μελέτη έδειξε το 2009 ότι ένας μήνας σπουδών στην Αλοδαπή μειώνει κατά 5% την πιθανότητα παραμονή σε μια χώρα για εργασία. Και μάλιστα η σχετική μελέτη της Ολλανδίας φανταστείτε τι αποτελέσματα θα είχε αν γινόταν στη Γαλλία ή στην Ελλάδα δεδομένου του ποσοστού ανεργίας των νέων. Πρόκειται για ένα φαύλο κύκλο. Γιατί όταν επενδύουμε στην ανώτατη εκπαίδευση ε, και ουσιαστικά εξυπηρετούμε τις πιο εύπορες χώρες και όχι τους ε, νέους πτυχιούχους, γιατί μερικοί από αυτούς ε, θα πάνε στην Αλοδαπή και θα απασχοληθούν σε λιγότερο ειδικευμένες εργασίες από αυτές που κανονικά θα δικαιούνταν λόγω βάση πτυχίου. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόβλημα για να μην ενισχύσουμε τις ήδη μαζικές, μαζικές ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μέλων. Ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε τον κύριο Οφλίν. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με πολλά από τα σχόλια που ακούσαμε και μάλιστα ε, μερικές φορές θα πρέπει να είμαστε πιο ριζοσπαστικοί γιατί αν η ε, Ευρωζώνη ακολουθήσει μία ε, φεντεραλιστική πορεία θα πρέπει να γίνει μια, μεταφο... μια ένωση των μεταφορών. Να δούμε τις οικονομικές διαφορές μεταξύ Γερμανίας και Ιταλίας από, την... Ε, από τον αρχικό σχεδιασμό. Θα πρέπει κάπως ε, να αντιδράσουμε ή να αλλάξουμε ριζικά το σύστημα ή θα γίνουμε μάρτυρες αυτών των, των μαζικών μετατοπίσεων και μετακινήσεων. Στην Ιταλία, Γερμανία, βλέπουμε ότι στην Ιταλία οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί θα γίνουν οι βασικοί χρηματοδότες μιας ένωσης των μεταφορών, των ευασμάτων, γιατί ε, στις χώρες του Νότου δεν θα έχουν καμία προοπτική ε, οι νέοι, αλλά αν θέλουμε οι νότιες χώρες να, να αναπτύξουν την παραγωγικότητά τους ε, και να πλησιάσουν προς το μέσο όρο της Ευρωζώνης, τότε θα χρειαστούν πολύ σημαντικές επενδύσεις στην παιδεία και την κατάρτιση. Αυτό θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών. Αυτό είναι το κατάλληλο μήνυμα και όχι ένα μήνυμα απόγνωση. Βέβαια κάτι τέτοιο θα είναι δαπανηρό και σίγουρα τα Υπουργεία Οικονομικών δεν έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν μια τέτοια προσπάθεια. Αν η Ευρωζώνη συνεχιστεί θα πρέπει να γίνει μια συνολική ε, ένωση των μεταφορών και οι βόρειες χώρες που έχουν ε, εποφεληθεί από το ευρώ και έχουν σχετικά χαμηλές ισοτιμίες θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν τις νότιες χώρες που δυστυχώς η οικονομία τους έχει χάσει σημαντικά σε ανταγωνιστικότητα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η Julie Βόλτ. Δύο λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ. Με προβλημάτισε η πρόταση της κυρίας Μπιλτ ότι προγράμματα σαν το Erasmus Plus δημιουργούν πρόβλημα για τους νέους που προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας ή να ακολουθήσουν μια κατάρτιση. Κυρία Μπίλτ, για τη δική σας παρέμβαση μιλάω. Δεν με ακούτε. Σχολιάζω τις δικές σας παρατηρήσεις περιπτώσει, ξαναρχίζω. Με προβλημάτισε το σχόλιο σας ότι το πρόγραμμα Erasmus Plus ήταν ένα από τα προβλήματα για τους νέους που προσπαθούν να βρουν μια θέση εργασίας ή ένα πρόγραμμα κατάρτιση. Το περασμένο Σαββατοκύριακο ήμασταν με τη Σιλβή Γιγιόμ στο, στην Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για του νέου, από 9.000 νέοι από όλη την Ευρώπη, νέοι που πιστεύουν στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο και Όραμα, ε, ήταν σαφής πιστεύουν ότι το Erasmus Plus είναι πραγματικά πολύ σημαντικό σχέδιο νευραλγικής σημασίας για, την, για το διαπολιτισμικό διάλογο, για την απόκτηση δεξιοτήτων που θα τους επιτρέψουν να χτίσουν τη δική τους επιχείρηση ή να βρουν μια θέση απασχόλησης. Αυτό είναι το αίτημα των νέων και οι νέοι θέλουν την κινητικότητα, θέλουν το Erasmus γιατί έτσι έχουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν ανά την Ευρώπη, ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση και πέραν του συνόρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συναντηθούν, να ονειρευτούν, να σχεδιάσουν νέα προγράμματα και σχέδια και να φτιάξουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Νομίζω ότι και η Επιτροπή μας συμφωνεί ότι το Erasmus Plus είναι ένα αξιόλογο ευρωπαϊκό πρόγραμμα και αξίζει υποστήριξης. Και δεν είναι μόνο τα εύπορα παιδιά που θα σπουδάσουν σε πανεπιστήμια σε άλλες χώρες. Το, το συν του έρασμος είναι ότι άλλα προηγούμενα προγράμματα όπως η νέη ενδράση, γιατί αυτό το πρόγραμμα νέη ενδράση ε, κατευθυνόταν και είχε δικαιούχους τους πιο ευάλωτους νέους με δυσλεξία, με μαθησιακές δυσκολίες, με αυτισμό και το γνωρίζω από πρώτο χέρι, γιατί πριν ασχοληθώ με την πολιτική, με αυτά τα θέματα ασχολούμαι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να στραφώ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Θέλετε να... Α, είστε εδώ. Παρακαλώ, δύο λεπτά εσείς. Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση για την, για την απασχόληση, κοινωνικά θέματα και την κοινωνική ένταξη. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα τα θέματα που πραγματεύεται αυτή η γνωμοδότηση. Οι επενδύσει στην παιδεία, στην κατάρτιση, σε ποιητική, ε, ε, ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, ε, σε συνδυασμό με τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Και πραγματικά θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη θέση στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στις ειδικέ συστάσεις αναχώρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Μαΐου. Οπότε δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάπτυξη αυτή τη πρωτοβουλία και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον εισηγητή και τους κοιόδη εισηγητές για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τέλο. Να δώσω το λόγο και πάλι στον ε, συντάκτη γνωμοδότησή μα τον κύριο Χουντή, αν θέλει να κάνει παρατηρήσει. Παρακαλώ, κύριε Χουντή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες απόψεις που κατέθεσαν ε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας εξομολογηθώ ότι ξέρω τη δυσκολία του θέματος. Διότι και από τις τοποθετήσεις σας, όσο αφορά το ποια είναι η εικόνα και ποια είναι η κατάσταση σήμερα στο τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης, νομίζω ότι συμφωνούμε. Και όπου δεν συμφωνούμε έρχονται τα στοιχεία, τα οποία αξιοποίησα, τα στοιχεία της Eurostat, που μιλάει για αυτά τα φαινόμενα τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα και οικοδομείται η γνωμοδότηση. Το δεύτερο στη συζήτηση και θα δεχτώ και βεβαίως και η συζήτηση της τροπολογίας είναι οι αιτίε και τι μπορούμε να κάνουμε. Σας μιλώ πάλι ειλικρινά θα καταβάλω κάθε προσπάθεια να βρω κοινού τόπους γιατί όσο αφορά το πού οφείλονται και πώς μπορούν να θεραπευτούν αυτά τα προβλήματα τα οποία θίγει η γνωμοδότηση φοβάμαι ότι δεν έχουμε ίσως κοινή αντίληψη. Α, να σας πω ένα παράδειγμα. Όλοι μιλάμε ότι χρειάζεται χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης. Όμως γνωρίζουμε ότι μέσω της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου ο έλεγχος που γίνεται στους προπολογισμούς των κρατών μελών γίνεται με βάση την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Δηλαδή κάποιο κράτος που θα θελήσει να δώσει δαπάνες για την παιδεία θα κατηγορηθεί ότι πάει και ξεφεύγει το έλλειμμά του. Είναι αυτό που έχουμε ζήσει. Εκεί είναι οι αντιφάσεις τις οποίες προσπαθούμε και προσπαθώ και θα προσπαθήσω να τις ξεπεράσουμε για να τοποθετηθούμε σε θετικές προτάσεις. Θετικές προτάσεις. Και βεβαίως δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Ε, θα πάρουμε τις τροπολογίες, θα καταθέσει τις τροπολογίες και σας ξαναλέω θα κάνω σοβαρή προσπάθεια προκειμένου να βρούμε κοινό τόπο ούτως ώστε να διατυπωθούν οι δικέ μα εκτιμήσει και προτάσει που να μπουν στην έκθεση απασχόληση για να πιέσουν την Κομισιόν στο πλαίσιο όλων αυτών των συζητήσεων να πάρει καλύτερε, θετικότερε κατευθύνσει όσον αφορά τα ζητήματα που στο τέλο τέλο είναι και ο πυρήνα και η ουσία τη Επιτροπή μα <laughs> όλο αυτό το διάστημα, όπω ε, τουλάχιστον το αντελήφθη και επομένω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και του συναδέλφου για τι παρατηρήσει. Ε, περιμένω τι ε, τροπολογίε, το χρονοδιάγραμμα το θέσατε εσεί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Ευχαριστώ. Ja, vielen herzlichen Dank. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, δεν βλέπω πολύ καλά ποιος είναι εδώ για αυτήν την αίθουσα. Και πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, είχε στήσει το λόγο πάλι η κυρία Μπίλντ, την οποία δεν την είδα. Σας παρακαλώ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν πειράζει. Να απαντήσω στην κυρία Ward, η οποία μάλλον παρανόησε λίγο τα λόγια μου. Και εγώ την Κυριακή πήγα να συναντήσω τους νέους, διότι ε, είχα και εγώ μια ομάδα εκεί. Και ίσα ίσα που πιστεύω ότι το Εράσμους ε, και πολύ καλό είναι και έχει λειτουργήσει πολύ καλά ως τώρα. Απλώς έλεγα να προσέξουμε ώστε το Εράσμος που ανοίγει σε πολλά πράγματα τους ορίζοντες να μην συμβάλλει στην φυγή των ταλέντων από τον Νότο και την φυγή γενικότερα από την Ευρώπη ε, με τόση ποικιλία στις γλώσσες και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ. Προθεσμία για τροπολογίες, επαναλαμβάνω, 12 Ιουνίου, 11 η ώρα και ψηφοφορία στην τελευταία μας συνεδρίαση πριν τις καλοκαιρινές διακοπές, 11 Ιουλίου. Σας εύχομαι επιτυχία στην περαιτέρω εργασία και συζήτηση και είμαι πεπισμένη ότι θα καταλήξουμε σε ευρεία συνένεση εδώ στην Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε τα θέματά μας στις αρμόδιες επιτροπές. Περνάμε στο 7 τώρα. Είναι ενημέρωση για την ε, συνεδρίαση της ομάδας παρακολούθησης ε, του Brexit της Κούλτ και να δώσω το λόγο πρώτα απ' όλα στον κύριο στο Ιεύσκι για να μας παρουσιάσει τις τελευταίες εξελίξεις. Έχετε το λόγο κύριε Στρογεύσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Ε, θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός. Καταρχήν, από τη μία πλευρά έχουμε το επίσημο έγγραφο και έχετε διαπιστώσει από το έγγραφο αυτό σε ποια φάση βρίσκονται οι διαπραγματεύσει ό,τι αφορά την αποχώρηση τη Μεγάλη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα οι διαπραγματεύσει επισπεύστηκαν τον τελευταίο καιρό και από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ε, μάλλον θα έχουμε ένα είδος εταιρικής σχέσης αλλά και μια μεταβατική περίοδο και όλα δείχνουν ότι ως προς τα θέματα των δικών μας ενδιαφερόντων, δηλαδή ε, το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί μετά την ε, μεταβατική, όπως λέμε, περίοδο. Καταρχήν, κάποια πραγματικά περιστατικά. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτησε το ψήφισμα για τους βασικούς όρους της μελλοντικής σχέσης, ε, εταιρικής σχέσης. Έγινε αυτό το Μάρτιο στο Στρασβούργο φέτος. Για πρώτη φορά μας ζητήθηκε να μιλήσουμε για ε, τη μία πιθανή ε, σύσταση ε, Επιτροπής Παρακολούθησης που υπέβαλε συστάσεις που λύθησαν υπόψη στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά την φάση αυτή προβλέπω ότι το φθινόπωρο δεν θα μας ξαναζητηθεί να αποφαθούμε για θέματα που ήδη αναφέραμε στο ψήφισμά μας. Αλλά θα δούμε την αλληλουχία των φάσεων της διαπραγμάτευσης ε, και κυρίως μας ενδιαφέρουν τρεις τομείς. Καταρχήν το έρασμος πλάς, η αναγνωρισιμότητα των ε, διπλωμάτων, των τίτλων σπουδών και επίσης ε, μας ενδιαφέρουν τα θέματα των, των δικαιωμάτων των πολιτών. Και μάλιστα σε αυτή τη φάση δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτή μια συμφωνία σύνδεσης γιατί δεν έχει μείνει πολλούς χρόνους γι' αυτό. Η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλει ακόμη με σαφήνεια τη θέση της ε, και τις σκέψεις της για τις μελλοντικέ της σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, γιατί μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ό,τι αφορά τα δικά μας ε, ενδιαφέροντα. Καταρχήν, έχει ε, ε, επιτευχθεί συμφωνία ό,τι αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Και εδώ μπορούμε να έχουμε κάποιες εγγύσεις ότι τα επαγγελματικά, τα τυπικά επαγγελματικά προσόντα και μετά την ε, έξοδο αλλά και κατά τη μεταβατική περίοδο θα ε, γίνεται αναγνώριση. Και κατά την ε, παραμονή, μάλλον και κατά την μεταβατική περίοδο θα γίνεται αναγνώριση. Επίσης, τα προγράμματα Erasmus Plus, Δημιουργική Ευρώπη και Ευρώπη των Πολιτών θα συνεχιστούν αμετάβλητα και στη μεταβατική περίοδο, δηλαδή μέχρι το 2021. Στην ερώτηση που υπέβαλα εγώ, αν θα υπάρξει δυνατότητα παράτασης ε, της μεταβατικής περίοδου, μου απάντησαν καταφατικά. Ε, σε περίπτωση όμως ε, παράτασης της μεταβατικής περίοδου και αλλαγής της γνώμης του Ευρωπαίου αλλαγή τη γνώμη του Ηνωμένου Βασιλείου και επιθυμίες επαναφορά, θα πρέπει να ξεκινήσει όλη η διαδικασία ε, ένταξη, σαν να έχει εξέλθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παραμείνει στη Σύμβαση των Ευρωπαϊκών Σχολείων σίγουρα μέχρι το τέλο τη σχολική χρονιά 2020-2021. Τι θα γίνει μετά. Δυστυχώ, σήμερα δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε τι θα γίνει μετά την περίοδο αυτή. Και τέλος, ε, η συμφωνία της αποχώρησης ε, θεσπίζει μία μεταβατική περίοδο. Δεν θα ήταν όμως ε, χρήσιμο αν μέχρι τον επόμενο Απρίλιο είναι έτοιμη η σχετική συνθήκη, η συνθήκη αποχώρησης. Όλα όμως δείχνουν ότι δεν θα είναι έτοιμη, δεν θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η σύμβαση, η συμφωνία. Οπότε Κατά πάσα πιθανότητα, μέχρι το 2021 η το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι υποχρεωμένο να εφαρμόσει το κοινοτικό κεκτημένο μέχρι τότε. Θα αποτελεί τμήμα τη κοινή αγορά, τη Θελωνιακή Ένωση και θα συμβάλλει στον κοινοτικό προπολογισμό. Επίση, θα υπόκειται στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Όμω, δεν θα συμμετέχει στη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Για προφανεί λόγου. Μπορούμε να σκεφτούμε ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα θέλει να παρατείνει τη μεταβατική της περίοδο επειδή δεν θα συμμετέχει κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τώρα, τι θα συμβεί μετά το 2021, μετά την λήξη της μεταβατικής περίοδου. Όλα αυτά θα, κανονικά θα πρέπει να τα περιέχει η Συμφωνία Σύνδεσης. Αλλά η εγγύηση συνέχιση των σημαντικών προγραμμάτων, το Erasmus Plus της Δημιουργικής Ευρώπης Ευρώπης των πολιτών, δεν ε, εξασφαλίζεται. Δεν υπάρχει εγγύηση για τη συνέχιση μετά την ε, λήξη της μεταβατικής περίοδου. Σε ό,τι αφορά τις ε, εξετάσεις και το απολυτήριο ηλικίου. Όσοι θα λάβουν το απολυτήριό του μέχρι το 2020 μπορούν να είναι ήσυχοι ότι τα απολυτήριά του θα αναγνωριστούν. Βέβαια, μετά το 2021 δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τίποτα για το κατά πόσο θα γίνεται αναγνώριση των απολυτήριων. Αυτά, κυρία Πρόεδρε, ήμουν αλακωνικός. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Σδρογεύσκη. Ευχαριστούμε για τα πορίσματα αυτά τη ομάδα παρακολούθηση. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ τις εξελίξεις. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικά μας ενδιαφέροντα και τις δικές μας αρμοδιότητες. Και στη διάσκεψη Πρόεδρων Επιτροπών είμαι σίγουρη ότι θα επανέλθουμε στο ζήτημα αυτό. Και φυσικά θα σας κρατώ ενήμερους για τα όσα θα υποθούν στην ε, διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών. Δεν θα κάνει το λόγο. Ή μάλλον ο κύριος Φλίν, για ένα λεπτό. Εδώ δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, φαίνεται. Ε, ο, η Βρετανή Πρωθυπουργό φαίνεται ότι θα κάνει ό,τι λένε ο κύριος Μπαρνιά και η υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν ε, φύγουμε από το backstop και την Τελωνιακή Ένωση και την Ενία αγορά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή και η Ιρλανδία λένε ότι το ζήτημα των συνόρων δεν έχει λυθεί και ότι μόνο τότε θα μπορεί να φύγει από την Τελωνική Ένωση και την Ενία Αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, ο Πρωθυπουργό μα όμω ε, είναι πρόθυμη να υπογράψει επιταγέ και να ευχαριστήσει για τι οικονομικέ ε, απαιτήσει. Εφόσον λοιπόν ελέγχει το Ηνωμένο Βασίλειο η Πρωθυπουργό αυτή και ε, όλη μας την πολιτική θα ε, ακολουθεί κάποιες φορές την, ε, τα όσα προτιμούν εδώ όσοι βρισκόνται σε αυτή την αίθουσα και γενικώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι μάλλον δυσάρεστο για μένα και το Βρετανικό λαό. Κάτι που δεν έχει φέρει σε καθόλου καλή θέση σήμερα το Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλος το λόγο. Οπότε είναι ένα θέμα που θα το ξαναδούμε. Και... Ευχαριστώ τον κύριο Στρογεύσκη και την ομάδα του για την εργασία της. Θα παρακολουθήσουμε με προσοχή το θέμα και περαιτέρω και ενδεχομένως θα επανέλθουμε. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημέρης της διάταξης. Είναι η μελέτη του Τμήματος Πολιτικής για τα, ταμεία, τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία επενδύσεων στον τομέα του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Θα θυμάστε ότι την ε, έκθεση αυτή την έχουμε παραγγείλει εδώ και καιρό γιατί είμαστε ενώπιον του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου και θέλουμε να αγωνιστούμε ότι τα θέματα των επενδύσεων για την εκπαίδευση για τον πολιτισμό θα παίξουν έναν ιδιαίτερο ρόλο. Και από το τόσο μεγάλο ποσό που χρηματοδοτούν τα κράτη-μέλη να αποδοθεί ένα ποσό και σε αυτούς τους τομείς. Όπως ξέρετε, τα διευθυντικά ταμεία τα διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη. Δημιουργήσαμε τη δυνατότητα, λοιπόν, να ζητήσουμε αυτά τα ποσά και θα ήθελα να... θα θέλαμε να ξέρουμε εάν τα κράτη-μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τα μέσα που τους δίνουν οι κανονισμοί για τα ταμεία ΕΣΥΦ για να υπάρξουν οι αναγκαίες επενδύσεις και για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Δηλαδή να τα αξιοποιήσουν όπως θέλουμε, όπως θεωρήσαμε και είναι λοιπόν πολύ επίκαιρη αυτή η έκθεση. Γιατί ξεκινάει ζήτηση για όλα τα νέα προγράμματα και θα λάβουμε θέση και για τα, τα διαφορετικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής και γενικότερα για τα ταμεία ΕΣΥΦ και γι' αυτό καλωσορίζω ιδιαίτερα τον Μάικ Κόιν και τον Μάλιν Κάτσμπεργκ από το Κέντρο για την ε, Στρατηγική και την Αξιολόγηση οι οποίοι κατήρτισαν αυτή την έκθεση με βάση την εντολή του τμήματος πολιτικής μας. Τους παρακαλώ να μας παρουσιάσουν τα αποτελέσματα. Ξέρω πως ήταν ιδιαίτερα αναλυτική μελέτη, την έχω ήδη διαβάσει και σας συστήνω να τη διαβάσετε όλοι, αλλά σας παρακαλώ να περιοριστείτε στα βασικά σημεία και ο καθένας σας θα έχει πέντε λεπτά για να μας παρουσιάζει τα αποτελέσματα, για να έχουμε και λίγο χρόνο για περαιτέρω ερωτήσεις και συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και σας δίνω το λόγο κύριε Κόιν ή όποιος θέλει από τους δυο σας να ξεκινήσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Να περάσω απευθείας στη μελέτη που εκπονήσαμε για τη χρήση των διευθυντικών και επενδυτικών κονδυλίων στον τομέα της εκπαίδευσης, παιδείας, αθλητισμού και νεολαίας. Εξαιτία τη διάρθρωση τη έκθεση, πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στο νομικό πλαίσιο, του κανόνε βάσει των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια, έσυφο όπω τα έχουμε ονομάσει, έπειτα το βαθμό ε, στον οποίο πραγματικά προσφέρθηκε στήριξη για αυτού του τέσσερι μετά θα κάνουμε μια επισκόπηση των βασικών πορισμάτων και μετά θα δούμε τις επιπτώσει ε, όπως προβλέπονται για το μέλλον, με κάποιε συστάσεις μαζί. Ω προ το πλαίσιο λοιπόν που καθόρισε το τι μπορούν να προσφέρουν και σε τι μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια ΕΣΥΦ, οι, βασικότερες, οι βασικότεροι παράγοντε ήταν πρώτα απ' όλα όσο προβλέπει συνθήκη και μετά η περίοδο προγραμματισμού. Οι κανόνε, έσυφ δηλαδή. Στην τωρινή περίοδο, ε, την τρέχουσα περίοδο, βρήκαμε ότι η εκπαίδευση και η παιδεία έχουν μία παρουσία εξέχουσα. Μία από τις, από τους 11 θεματικούς στόχους που ε, έπρεπε να οργανώσει, οργανώσει ε, τις δαπάνες των 100 μελών ως στόχος. Όμως, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός δεν μπορούν να υποστηριχθούν αυτή καθεαυτή βάση των κονδυλίων ΕΣΥΦ, μόνο στα πλαίσια της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Έχουν λοιπόν άλλο καθεστώς. Και η νεολαία είναι ένας μείζον στόχος, κυρίως μέσω της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, Κάτι που είναι όμως εκτός ε, της δικής μας θεματικής και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε μόνο κάποια σχόλια. Ως προς τους κανόνες σημειώνουμε ότι υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί στην τρέχουσα περίοδο. Κυρίως λόγω της ε, θεματικής συγκέντρωσης που προβλέπει ότι τα κρατημέλη πρέπει να συγκεντρώσουν τις δαπάνες τους ε, σε τέσσερις μείζονες τομεί, όπως αναφέρονται στους στόχους, την έρευνα και την καινοτομία κυρίως, την στήριξη ε, στις, την πληροφορική, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ε, οικολογική οικονομία. Επίσης, για την εξάντε θα πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο πλαίσιο, λένε οι κανόνε, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να προβλέψουν έργα σε συγκεκριμένου τομείς. Λόγω χάρη η ευθύης ε, εξειδίκευση μπορεί να είναι μια προϋπόθεση για τις δαπάνες, την κοινοτομία και την έρευνα. Αυτό λοιπόν είναι το πλαίσιο. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να μεταφραστούν και να λειτουργήσουν σε εθνικό επίπεδο. Πολλές φορές μέσω συμφωνίας εταιρικής σχέσης, βάσει της οποίας οι προτεραιότητες των κρατών μελών καθορίζονται και επιλέγουν από το συνολικό πλαίσιο και έπειτα αυτά πρέπει να μεταφραστούν και σε επιχειρησιακά προγράμματα προγράμματα που περιλαμβάνουν συγκεκριμένε λεπτομέρειε για το πώ πρέπει να ε, διενεργηθούν διάφορε δαπάνε στα κράτη-μέλη. Και μετά καταλήγουμε στα συγκεκριμένα προγράμματα, τα έργα δηλαδή επιτόπου. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Για το γκρουπούσκουλο που βρίσκεται στην είσοδο της αίθουσας. Παρακαλώ, αποχωρήστε. Αν θέλετε να συζητήσετε, αλλά όχι μέσα στην αίθουσα, ενοχλείτε πολύ. Με συγχωρείτε. Μια γραφική παράσταση για να δείτε τις σχέσεις αυτές με προγράμματα όπου πραγματικά υπάρχει δράση και τα οποία επιλέγονται και καθορίζονται μέσω συμφωνιών σε εθνικό επίπεδο, δημόσιο και δυτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τους 11 θεματικούς στόχους και τις λεπτομερέστερες προτεραιότητες επενδύσεων και τα συνδυάζουν βεβαίως με την εξάρτητα αιρεσιμότητα για να προκύψουν τα αποτελέσματα. Εδώ παίζει το ρόλο της θεματικής συγκέντρωσης που σας έλεγα. Εντός λοιπόν αυτού του πλαισίου μελετήσαμε κατά πρώτον το τι πληροφορίες διαθέτουμε για τις δαπάνες, ιδίως στην τρέχουσα περίοδο. Και υπάρχουν δύο τρόποι να το εξετάσει κανείς αυτό. Πρώτα απ' όλα από τα πάνω προς τα κάτω, κοιτάζοντα τι πληροφορίες δημοσιεύονται από την Γενική Διεύθυνση Ρέτζιου. Και εδώ βρήκαμε λίγο την εκπαίδευση και η ε, κατάρτιση φτάνουν τα 39,2 δις ευρώ σε δαπάνες για την τρέχουσα περίοδο. Με βέβαια υπάρχουν και κάποιες ε, υπόγειες δαπάνες, θα τις έλεγα, που βρίσκονται σε άλλα κεφάλαια. Εδώ η εκπαίδευση και η κατάρτιση λόγου χάρη φαίνεται να είναι πολύ σημαντικές ως μέσα για να πετύχουμε άλλους στόχους. Οι περισσότερες δαπάνες στον αθλητισμό και τον πολιτισμό βρίσκονται σε άλλα κεφάλαια. Ο αθλητισμός λοιπόν και η παιδεία ο πολιτισμός μάλλον, χρησιμοποιούνται ακριβώς ως μέσα, ως οχήματα θα λέγαμε, για να πετύχουμε άλλους στόχους. Για τους ε, συνολικούς αριθμούς, δεν είναι πολύ σαφές το τι γίνεται με τις δαπάνες χώρους κρατικού συμφέροντος. Γι' αυτό δεν μελετήσαμε αυτή τη διάσταση, αλλά τις επιτόπου πληροφορίες που μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε. Με οκτώ κράτη-μέλη, τα βλέπετε στη διαφάνεια ποια ήταν, και Παρατηρήσαμε το τι συμβαίνει επί τόπου με συγκεκριμένα προγράμματα και το βαθμό κατά τον οποίο ε, εξυπηρετούνταν συγκεκριμένοι τομεί προτεραιότητα σε αυτά τα προγράμματα. Ωστόσο, είναι πολύ διαφορετικέ πληροφορίε που δημοσιοποιούν τα διάφορα κράτη-μέλη ανάλογα και τι, και τι λεπτομέρειε ε, αποκαλύπτουν. Σε κάποια κράτη-μέλη βρήκαμε πολλά στοιχεία, σε κάποια άλλα όχι. Ε, τα βασικά μα πορίσματα, πολύ σύντομα. Η εκπαίδευση, την κατάρτιση βρίσκονται παντού και ως στόχοι πολλές φορές, αλλά και ως ένα μέσο να επιτευχθούν άλλοι στόχοι. Για παράδειγμα, εάν κανείς προσπαθεί να προωθήσει τη, μια τεχνολογία πληροφορίας, πολλές φορές αυτό ε, καταχωρείται ως ε, κατάρτιση. Ε, και βρίσκονται και σε άλλα κεφάλαια, όπως έλεγα προηγουμένως. Η Ιταλία που έχει ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για τον πολιτισμό και η Πολωνία που δίνει μεγάλη έμφαση στον πολιτισμό είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Αλλά άλλε χώρε δεν κάνουν το ίδιο. Ιδίω ε, στι προηγούμενε περιόδου και την τρέχουσα. Η ευφυή εξειδίκευση πολλέ φορέ έχει να κάνει με τον πολιτισμό και, την, ε, και το χώρο της δημιουργίας καθώς και τον αθλητισμό. Αυτοί είναι τομεί που μα ενδιαφέρουν. Αλλά ο αθλητισμό γενικώ δεν έχει τόσο μεγάλη προβολή ω στόχο. Όμω, ε, προκύπτει παντού. Υπάρχουν δραστηριότητε αθλητικέ, πολύ συχνά που στόχο έχουν να επιτευχθεί μέσω αυτών άλλο στόχο. Παρόλο που δεν είναι τελείω ξεκάθαρο, ε, θεωρούμε ότι υπήρξε μείωση στην τρέχουσα περίοδο των δαπανών για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Ε, λόγω της θεματικής συγκέντρωσης. Μόνο μια-δυο χώρες μας έδωσαν στοιχεία όπου συνέβαινε κάτι διαφορετικό. Η νεολαία είναι ένα σημαντικό θέμα παντού, ιδίως όμως στις χώρες με υψηλή ενεργεία των νέων, όπως για παράδειγμα στην Ισπανία και την Ιταλία. Επίσης, δυο, τρεις, ίσως και τέσσερις τομείς συνδυάζονται ε, σε κάποιο πρόγραμμα με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό μαζί, ας πούμε, για τους νέους αλλά υπάρχουν και σημαντικές ε, σχέσεις αλληλεπίδρασης με το Erasmus in και την Δημιουργική Ευρώπη, κυρίως γιατί το Erasmus in έχει δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική ε, συνιστόσα. Τώρα, οι επιπτώσεις για το μέλλον. Για να το μελετήσουμε αυτό προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε κάποια κοινά θέματα σε όλους τους τομείς που μελετήσαμε και ήταν σαφέ ότι και στους τέσσερις αυτούς τομείς έχουμε να κάνουμε με την ανθρώπινη διάσταση σε αντιδιαστολή με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ανθρώπινη λοιπόν διάσταση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης είναι πολύ χαρακτηριστική στους τέσσερις τομείς που μελετούμε. Οι τομείς αυτοί ενθαρρύνουν με διαφορετικό τρόπο την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων, τη δημιουργικότητα, την αφοσίωση και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Είναι λοιπόν σοβαροί παράγοντες είναι οι τομείς αυτοί οι σοβαροί παράγοντες που διευκολύνουν και καλλιεργούν την ανάπτυξη. Είναι το αντίβαρο, θα έλεγε κανείς, των παραγόντων που ε, καλλιεργεί τεχνολογική ανάπτυξη. Βέβαια, δεν έχουν ακόμη τόσο μεγάλη προβολή στα πλαίσια των κονδυλίων ΕΣΥΦ. Παρόλο που είναι αυξανόμενη ε, σημασία από απ' όλα λόγω του διεθνού ανταγωνισμού ούτω ή άλλω, αλλά και τη αυτοματοποίηση η ανθρώπινη δραστηριότητα, η ανθρώπινη συμβολή εδώ θα αρχίσει να γίνεται ολοένα και πιο σημαντική, καθώ κάποιε θέσει εργασία την καθιστώνται από μηχανήματα και ρομπότ. Ο δρόμο για το μέλλον, λοιπόν. Αυτό που μας απασχόλησε ήταν οι δυνατότητες να βρούμε ξεχωριστά επιχειρήματα για να στηρίξουμε τον καθέναν από αυτούς τους τέσσερις τομείς ξεχωριστά. Αυτό όμω είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να βρει κανεί ε, επιχειρήματα υπέρ ενό συγκεκριμένου τομέα στο πλαίσιο των δαπανών ΕΣΥΦ. Γι' αυτό προτείνουμε μια συνολικότερη προσέγγιση. Συνολικότερη προσέγγιση που θα μπορούσε να έχει και περισσότερη επιρροή και επίδραση μακροπρόθεσμα. Ως προς τις συστάσεις μας λοιπόν, ακόμα απομένουν πολλά να γίνουν μόνο και μόνο για να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για τη σημασία των τεσσάρων αυτών τομέων. Ε, οι ευρωβουλευτέ εδώ μπορούν να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στι εκλογικέ του περιφέρειε, αλλά γενικότερα. Ε, κάτι άλλο που είναι σημαντικό να υποθεί μεταξύ των συστάσεων είναι ότι το μέλλον των δαπανών για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να έχουν ω κεντρικό θέμα την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων δεξιοτήτων και δυνατοτήτων. Αυτά θα γίνουν μοχλή για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει μια μνήμα στους τέσσερις αυτούς τομείς βεβαίως, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχύσουμε την παρουσία τους με τη χρήση αυτού του θέματος, αυτής της θεματικής, λόγω χάρη μεταξύ των κριτηρίων για την εξάντε ε, ρεσιμότητα. Επίσης, πρέπει να πλαισιώσουμε αυτήν την προσέγγιση ε, με, μια, ε, με ένα βλέμμα που να κοιτάζει προς το μέλλον θα πρέπει να έχουμε μια μακρόπνοη προσέγγιση, ε, ιδίως για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επίσης, μια σειρά από άλλους στόχους αναφέρονται μεταξύ των συστάσεων. Λόγου χάρη το να τονιστεί η σημασία του ρόλου της άτυπης εκπαίδευση και σε άλλου τομεί. Αυτοί μπορεί να είναι μηχανισμοί για να επιταχθούν άλλοι στόχοι όπως είπα, οπότε αν κανείς εξετάσει το πώ ε, χρησιμοποιούνται τα διεθνωτικά κονδύλια, ε, υπάρχει μεγάλη έμφαση στου στόχου και τα αποτελέσματα. Λιγότερο στο μέσο, στο μηχανισμό που επιτρέπουν να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα και στόχου. Αυτοί οι τέσσερι όμω τομεί είναι πολύ σημαντικοί ω μέρο του μηχανισμού για να πετύχουμε άλλου στόχου. Είναι σαν τα γρανάζια. Και γι' αυτό θα πρέπει να του δοθεί μεγαλύτερη προβολή. Θα πρέπει επίση να υπάρξει συγκεκριμένη παρουσίαση σε μοντέλα των, ε, προγραμ... των διαδικασιών με τι οποίε εφαρμόζονται τα προγράμματα μέσω του σχεδιασμού των προγραμμάτων, τη συλλογή στοιχείων για επιβολή εκθέσεων και τη αξιολόγηση. Η ευφυή εξειδίκευση θα πρέπει να συνεχίσει να αντικατοπτρίζει ακριβώς την ε, σημασία της ανθρώπινης διάστασης και βεβαίως να υπάρξει και κατάλληλη ε, το κατάλληλο σύστημα παρακολούθηση από τι αρχέ των κρατομελών για να παρακολουθούν τι ακριβώ συμβαίνει στην πράξη. Επίση, υπάρχουν πολλέ ε, οργανώσει ε, στον έξω κόσμο, ε, πολλέ ενώσει που είναι πολύ δραστήριε στον χώρο αυτό και πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτέ τι οργανώσει, αυτέ τι ενώσει, διότι πραγματικά ωφελούν όχι μόνο του εαυτού του, αλλά πρέπει να τους βοηθήσουμε να γίνουν ε, πιο επαγγελματικοί στην προσέγγιση τους, ώστε η οικονομική και η κοινωνική ανάπτυξη να έρθει και στα δικά τους χέρια. Ε, να ε, υποστηριχθούν στο δυνατόν περισσότερο, λοιπόν, για να συμβάλλουν. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με βάση τη διαδικασία ping-pong θα γίνεται μία ερώτηση και θα απαντάτε απευθείας. Ερώτηση-απάντηση. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει, αν δεν θέλει κανείς να ξεκινήσω εγώ. Να ξεκινήσω εγώ. Θεωρείτε λοιπόν ότι η δημιουργία δυνατοτήτων ούτως ώστε τα διαθροτικά ταμεία να μπορούν να αξιοποιηθούν και για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό. Θεωρείτε ότι συνολικά έχει επιτύχει. Θεωρείτε ότι τα κράτη-μέλη το γνωρίζουν αυτό. Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ότι μπορούν να την αξιοποιήσουν. Γιατί ξέρουμε ότι στον τομέα του πολιτισμού πολύ συχνά είναι αρμόδια η τοπική αυτοδιοίκηση. Και όπως ξέρετε όταν πρέπει να γίνουν οικονομίες ε, το πρώτο που κόβουμε είναι ο πολιτισμός. Γνωρίζουν λοιπόν ε, οι αρχές αυτές τι δυνατότητες ή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να γίνει ευρύτερα γνωστό και υπάρχουν ποσοστά για το ΕΣΥΦ πόσα προγράμματα συνολικά έχουν εκτελεστεί σε σχέση με άλλους τομείς. Δεν ξέρω αν μπορείτε να μου δώσετε ποσοστά, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον για μας. Απάντηση. Είναι πολύ δύσκολο να σας πω ακριβώς τι συμβαίνει. Επιτόπου. Όπως σας είπα, τα επίσημα στοιχεία τα παρουσιάζουν όλα με βάση τους γενικούς στόχους. Αν υπάρχει ένα πρόγραμμα για τον πολιτισμό ή τον αθλητισμό που αφορά την ε, εξέλιξη ε, τεχνολογίας πληροφόρησης θα εμφανίζεται ως τεχνολογία πληροφόρησης. Ο μόνος τρόπος να καταλάβουμε περί πρόκειται είναι να εξετάσουμε το κάθε ένα πρόγραμμα που είναι χιλιάδες χωριστά. Το επιχειρήσαμε σε έναν βαθμό, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές πρακτικές ε, για την ε, παρουσίαση της πληροφορίας. Για παράδειγμα, στη Δανία είναι πολύ καλά τα πράγματα. Φαίνεται γιατί ακριβώς έχει δαπανηθεί το κονδύλι για κάθε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά για τι μεγαλύτερε χώρε είναι πιο δύσκολο. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, υπάρχουν 64 επιχειρησιακά προγράμματα. Ορισμένα είναι εθνικά, ορισμένα είναι περιφερειακά. Είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσει τι ακριβώ συμβαίνει. Καμιά φορά οι περιφέρειες δημοσιεύουν στοιχεία, άλλες φορές εθνικές αρχές και είναι πραγματικά τεράστια προσπάθεια να καταλάβεις ε, τι γίνεται. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα δαπανώνται για αυτό το τομέα. Αλλά έχουμε κάνει και κάποιες μελέτες στο παρελθόν για τις δαπάνες των διαθροτικών ταμείων για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, όπου δίνουμε πολλά παραδείγματα. Και σαφές είναι ότι στους δύο τομείς αυτούς ε, υπάρχει πολλή δημιουργικότητα, πολλή εφευρετικότητα. Πολλά προγράμματα αξιοποιούν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και φυσικά και την εκπαίδευση και την κατάρτιση για να ε, προωθήσουν άλλους στόχους για παράδειγμα καινοτομία, τεχνολογία, ακόμη και κοινωνική συμμετοχή. Και αυτές οι προσπάθειες ε, φτάνουν σε πολύ συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού και επιτυγχάνουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Πολλά γίνονται λοιπόν. Αλλά ω τελικό σχόλιο είναι ότι θεωρούμε, χωρί να είμαστε απόλυτα σίγουροι, αλλά υπάρχουν αρκετά στοιχεία από αρκετέ χώρε ότι η θεματική συγκέντρωση έχει ως επίπτωση ότι δαπανώνται λιγότερα ιδιαίτερα για τον πολιτισμό και τον αθλητισμό από τις προηγούμενες ε, προγραμματικές περιόδους. Αλλά έχουμε μία πολύ μερική εικόνα. Ίσως λοιπόν να είναι λανθασμένη αυτή η εκτίμηση. Είμαστε λίγο διστακτικοί στο να εξαγάγουμε αυτό το συμπέρασμα. Ευχαριστώ πολύ, λέει Η Σύλβια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, διότι προφανώς μια αναγνώση δεν κάναμε στη μελέτη σας, αλλά πρέπει να γίνει και μια πιο εντελεχής μελέτη. Εδώ μας ενδιαφέρει σαφώς και το σκέλος on the field, το επιτόπου, που είναι αυτό που αφορά περισσότερο και το σύστημα, διότι τα δαπάνες είναι πολύ διαφορετικές στην Ιταλία. Το 90% των πόρων πάνε στα χέρια των περιφερειών. Καταλαβαίνω λοιπόν τη δυσκολία, γιατί και στην Ιταλία καταλαβαίνουμε πόσο το πλαίσιο που έχει γίνει ανοιχτών δεδομένων όπως λέγεται, open cohesion, ανοιχτή συνοχή, έχει διαμορφωθεί και είναι πολύ δύσκολο να αναγνωστεί σε κάποιες χώρες και το πώς διαχειρίζονται τους πόρους τους. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Στον ε, τωρινή μορφή του προγράμματος, του νέου προγράμματος για τη συνοχή και τα διευθυντικά ταμεία, πρέπει να κατανοήσουμε εάν το γεγονός ότι οι νέοι δείκτες για την ερμηνεία των προβληματικών καταστάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα κατά την κατάρτιση, αν η συμπερίληψη λοιπόν των δικτών αυτών μπορεί να δημιουργήσει κλίδες ανάγνωσης για το πού πάνε οι πόροι, πώς γίνονται οι δαπάνες, παύλα, πώς επιτεγκάνονται τα αποτελέσματα. Δηλαδή η εξάντε μα ε, μας αφορά ή θεματικές ε, ενότητες. Στην προηγούμενη περίοδο είχαμε κάνει μια μεγάλη μάχη για να περάσει ο όρος πολιτισμός στο στόχο 6. Το στόχο 6 που ήταν απλώς φυσική πόρη και προσθέσαμε και τους πολιτιστικούς. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Το πρόβλημα είναι ότι πρέπει όλα αυτά να γίνουν πιο ξεκάθαρα στις κλίδες ερμηνείας, ε, στους όρους ερμηνείας, εκ, της Πού είναι αυτό η οριζόντια ή θεματική κατεύθυνση. Ε, και κατά πόσον οι πολιτιστικοί πόροι πάνε, πώς να το πω τώρα, ε, πάνε εκεί που πρέπει και γίνονται πιο προφευλημένοι, ε, μπορούν να καταμετρηθούν. Και αυτό εξαρτάται και από το format, το μορφότυπο, το, τη μορφή που θα δώσουμε στην στους στόχους της πρότασης και κατά πόσο είναι συμβατή κατά την άποψή σας στα οριζόντια προγράμματα με τους ε, διευθυντικούς στόχους. Τα μεγάλα προγράμματα, το Erasmus η Δημιουργική Ευρώπη, αυτά πώς λειτουργήσαν στην πράξη κατά την άποψή σας. Είχαν μια αμοιβαία αναγνώριση ή ακολούθησαν ξεχωριστή πορεία. Διότι είδαμε ότι το σημειώσατε, υπάρχει χαμηλό επίπεδο συμπληρωματικότητα μεταξύ των κονδυλίων και τη στήριξη λόγω χάρη με τι υποτροφίε, τα όσα προσφέρει το Εράσμο κτλ. Είναι έτσι. Ξεκινάω από το τελευταίο σας σημείο. Όντως, άλλα προγράμματα όλο και περισσότερο συγκλίνουν με το ΕΔΕΤ, το Διαρθρωτικό και Επενδυτικό Ταμείο. Και αυτό ήταν και ο στόχος, η πρόθεση. Κάποια σχέδια που καθορίζονταν από το Erasmus Plus να αναλυθούν από το ΕΔΕΤ. Πάντως φαίνεται ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη σύγκληση για πολλά σχέδια και προγράμματα του Erasmus Plus και του Δημιουργική Ευρώπη αρχίζουν και ε, δίνουν έμφαση στα κοινωνικά αποτελέσματα. Κάτι που συνδέεται πιο φυσιολογικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Μακροπρόθεσμα, κατά τη γνώμη μας, ελοχεύει ο κίνδυνος με τη συγκέντρωση μόνο στα επίσημα πλαίσια που ναι μεν είναι πολύ σημαντικά αλλά όχι μόνο έμφαση σε αυτά. Όπως είπα και στην παρουσίαση στους τομείς που εξετάζουμε ε, διαπιστώνουμε ότι χρειάζονται μηχανισμοί ε, παροχής αποτελεσμάτων. Το είπα στην παιδεία και στην κατάρτιση που γίνεται φορέας για την υλοποίηση και άλλων αποτελεσμάτων. Γι' αυτό χρειάζεται η ανάπτυξη της παιδείας και της ανάπτυξης που θα χρησιμοποιηθούν για να υλοποιηθούν και αποτελέσματα. Η χρήση δηλαδή της παιδείας και της κατάρτισης για να παραχθούν αποτελέσματα και σε άλλους τομεί. Πάντως, για να έχουμε μια πλήρη επισκόπηση τη κατάστασης, δεν πρέπει να εξετάσουμε μόνο τους στόχους και τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τους δείκτε. γιατί αυτή ήταν η τάση που διαπιστώσαμε μέχρι στιγμής, επικέντρωση σε αυτά τα θέματα. Το θέμα είναι πώς θα περάσουμε και από του ε, διάμεσου μηχανισμού. Γιατί τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν ε, οι τρόποι αξιολόγηση που περάσαμε από τη θεωρία στην έμφαση που δίνουμε στους μηχανισμούς και, για να φτιάξουμε την αξιολόγηση. Οπότε δίνεται έμφαση στα τελευταία στοιχεία. Αλλά αυτό που λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου τομεί είναι η διαδικασία να προωθηθεί, γιατί έχουμε πολλές εξελίξεις, όχι μόνο στα θέματα παιδείας και κατάρτισης. Δώσαμε στη μελέτη και άλλα παραδείγματα με τον αθλητισμό, πώς χρησιμοποιείται ο αθλητισμός για να περάσουν κάποια, κάποια μηνύματα και για να έχουμε και επιστημονικές εξελίξεις μέσω της εμπλοκής και πιο περιθωριακών ομάδων και μάλιστα με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κοιτάω γύρω-γύρω. Έχει κανείς άλλες ερωτήσεις? Όχι. Α, α, παρακαλώ. Ο κύριος Γραμματικάκης. Βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα τη μελέτη και τον τρόπο που μας την παρουσιάσατε, παραδεχόμενος ταυτόχρονα πόσο δύσκολο είναι να βρει κανείς την πραγματική εικόνα πίσω από τα διαρθρωτικά προγράμματα. Εμένα ιδιαίτερα με ενδιαφέρει και εκεί σας παρακαλώ αν έχετε κάποιο σχόλιο το θέμα της ανεργίας των νέων που σύμφωνα με τα δικά σας στοιχεία εμφανίζει πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένες από τις χώρες της Ευρώπης ειδικά στην πατρίδα μου την Ελλάδα ενώ τα διαρθρωτικά ε, τα μία φαίνεται να απορροφώνται και μάλιστα κατά 100% μου έκανε εντύπωση αυτό από την άλλη η ανεργία φτάνει πολλές φορές και το 21%. Νομίζω για όλους μας, νομίζω για όλη την αίθουσα είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ανεργίας των νέων. Ξέρω ότι είναι δύσκολο το εγχείρημα να καταλάβει κανένας ακριβώς τι γίνεται πίσω από χιλιάδες επιγραφές, προγράμματα και χρήματα. Θα ήθελα λοιπόν εσείς αν έχετε κάποιο σχόλιο πάνω στο μέγιστο αυτό θέμα. Um, uh, Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το ΕΔΕΤ. Το τρόπος δηλαδή που τα κράτη-μέλη προσαρμόζουν το γενικό πλαίσιο στις επιμέρους περιστάσεις. Ε, εξετάσαμε πολλές χώρες, ε, όχι την Ελλάδα, αλλά στις 8 χώρες υπάρχουν μεγάλες διαφορές στην έμφαση που δίνουν στην ενέργεια γενικά και στην ενέργεια των νέων ειδικά. Στη Γερμανία και τη Δανία, για παράδειγμα, έχουμε την εντύπωση ότι δεν είναι ιδιαίτερο το πρόβλημα αυτό. Είναι θέμα περισσότερο ε, επανακατάρτισης ή κατάρτισης ε, εργαζομένων ή ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων. Εκεί δόθηκε η έμφαση περισσότερο στις χώρες αυτές. Ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία, για παράδειγμα, ε, ανεργία των νέων ήταν μείζον πρόβλημα και γι' αυτό φάνηκε στα επιχειρησιακά τους προγράμματα που έδωσαν περισσότερη έμφαση σε αυτό το θέμα. Οπότε είναι σημαντική ελαστικότητα που εξασφαλίζει το σύστημα για να προσαρμοστεί κάθε χώρα στις δικές της περιστάσεις. Ιδιαίτερα το θέμα της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων δεν ήταν τμήμα της, ε, το αντικειμένο της έκθεσης δεν μας ζητήθηκε να αγγίψουμε και σε αυτό το θέμα ειδικά. Εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο, αλλά όχι στην έκθεση. Πάντως, στις χώρες που υπάρχει πρόβλημα με το θέμα αυτό, υπάρχει μεγαλύτερη συμπληρωματικότητα με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Προσπαθούμε, προσπαθούν να συμμετέχουν, να μίξουν οι χώρες αυτές και νέους. Και προσπαθούν να αναπτύξουν τις δεξιότητε γενικώ του εργατικού δυναμικού. Πάντως η γενική μα εντύπωση είναι ότι φυσικά η νεολαία είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχει τη θέση της στο πρόγραμμα αλλά στη, στον πολιτισμό και στον αθλητισμό ε, εκεί είναι κάπως ορφανά αυτά τα θέματα γιατί ελάχιστα αναφέρονται ο ο αθλητισμός στα βασικά προγράμματα. Εκτός και αν προωθείται ειδικά από ένα κράτος μέλος. Είναι φτωχή συγγενής ουσιαστικά ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Αυτά, ευχαριστώ. Yeah. Ναι, ευχαριστώ πολύ εκ νέου. Τώρα πραγματικά δεν βλέπω κανένα άλλο θέλει το λόγο, οπότε σας ευχαριστώ θερμότατα για την παρουσίασή σας, για την παρουσίασή σας και φυσικά για τη μελέτη που εκπονήσατε που νομίζω ότι θα διαβάσουμε όλοι πολύ προσεκτικά γιατί αναφέρει σημαντικά στοιχεία για το πώς θα διαμορφώσουμε τα προγράμματά μας ε, καλύτερα στο μέλλον και θα μπορέσουμε, πιστεύω, να αξιοποιήσουμε καλύτερα τα διαδοτικά ταμεία. Και πέρα από την ανεργία των νέων, το οποίο βεβαίως αξιοποιεί ιδιαίτερα τους πόρους του κοινωνικού ταμείου. Αλλά και στον ε, τομέα της άτυπης κατάρτισης και στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Γιατί ξέρουμε ότι ο αθλητισμός έχει τεράστιο ρόλο για την ένταξη των νέων στην κοινωνία. Ιδιαίτερα για περιοχές μειονεκτικές. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Αυτά βεβαίως ε, σχετίζονται με τους στόχους και του Κοινωνικού Ταμείου και των Περιφερειακών Ταμείων. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε συγκεκριμένα πώς θα αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα αυτές τις δυνατότητες. Με πιο, πολύ πιο λειτουργικό τρόπο για τα ίδια τα κράτη-μέλη. Ούτως ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν προγράμματα που να αξιοποιούν αυτούς τους πόρους. Σας ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας και για την παρουσία σας. Και την παρουσίασή σας. Και σας εύχομαι καλή μέρα. Οπότε θα μπορούσαμε να περάσουμε στο 8 λέει η πρόεδρος αλλά η κυρία Σίγκαν η διευθύντρια της ε, DG Home είναι εδώ. Das sieht offensichtlich nicht so aus. Αλλά δεν είναι εδώ. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Θα μπορούσα να πάω και λιγάκι, ξέρετε εκεί που πηγαίνει κανείς. Λοιπόν, 10 λεπτά διακοπή και η κυρία Σιγκάν ελπίζω να έρθει λίγο νωρίτερα. Ούτως ώστε να μπορέσουμε να τελειώσουμε και νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ.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

Liebe... Αγαπητοί συνάδελφοι. Σίλβια. Liebe... Αγαπητοί συνάδελφοι. Περνάμε στο σημείο 9 της το πρόγραμμα ε, Ευρώπη για τους πολίτες και συζήτηση με την Κομισιόν για το επόμενο πρόγραμμα. Χαίρομαι που έχουμε μαζί μας την ε, κυρία Σιγκάν, Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Home. Νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που έρχεστε στην Επιτροπή μας, γιατί δεν έχετε αναλάβει εδώ και πολύ καιρό. Οπότε καλώς ήρθατε στην πρεμιέρα σας ενώπιον της Επιτροπής ε, Πολιτισμού, όπως γνωρίζετε όλοι στο τέλος Μαΐου είχαμε την πρόταση για το νέο προγράμματα αξίες και δικαιώματα των πολιτών. Είναι λοιπόν ε, σαφές τι προτίθεται να κάνει με το δικό μας εντό αγωγικών πρόγραμμα η Ευρώπη για τους πολίτες. Δηλαδή να το συνδυάσει με το υπάρχον πρόγραμμα δικαιώματα, ισότητα και ηθαγένεια της Ένωσης. θέλει να απλουστεύσει η Κομισιόν τα προγράμματα αυτά. Οπότε είναι κάτι το καλοδεχούμενο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι αποδυναμώνεται το κείμενο επίσης. Και η ουσία του προγράμματος σε μεγάλο βαθμό ε, έχει λιγότερα καθήκοντα. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτό είναι πρόβλημα αυτό εξαρτάται από το τι θα γίνει για την περαιτέρω εφαρμογή του προγράμματος και για τους συγκεκριμένους στόχους της. Όπω είναι τώρα τα πράγματα, τα ετήσια προγράμματα πρέπει να εγκρίνονται μέσω ε, εφαρμοστικών και όχι κατεξοδότηση πράξεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το συζητήσουμε περαιτέρω. Όπως και το θέμα της πρικοδότησης των προγραμμάτων. Βεβαίως είμαστε στην ευνοϊκή κατάσταση ότι αντίθετα με το προηγούμενο πρόγραμμα όπου είχαμε επιλέξει ή χρειάστηκε να επιλέξουμε νομική βάση για την Κομισιόν είχαμε επιλέξει μια νομοθετική βάση που δεν μας έδινε σχεδόν καμία δυνατότητα να συμμετάσχουμε. Τώρα όμως είμαστε στην πολύ πιο ευχάριστη θέση ότι βρέθηκε μια άλλη λύση και εμείς ως Κοινοβούλιο επιτέλους μπορούμε να έχουμε πλήρες δικαίωμα διαμόρφωση του προγράμματος. Και από ό,τι φαίνεται θα υπάρξουν και περισσότερα κονδύλια, τουλάχιστον από πρώτη άποψη. Έτσι φαίνεται. Αλλά εάν εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα το προϋπολογισμό για τον τομέα της ηθαγένειας, για τη συμμετοχή προβλέπονται 232 εκατομμύρια. Αλλά τα 188 είναι από το παλιό πρόγραμμα. Μεταφέρονται δηλαδή και μόνο 45 εκατομμύρια από την Τέγκε Γιούστ θα αφιερωθούν για τα θεμελιώδη δικαιώματα και κοινωνία των πολιτών. Οπότε καθίστατε σαφές ότι για, τα, για τους στόχους του παλιού προγράμματος για την Ιθαγένεια δεν θα υπάρξουν επιπλέον πιστώσεις. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε. Γιατί όλοι ως βουλευτές τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πάντα το πρόβλημα ότι διάφοροι δήμαρχοι απευθύνονταν σε μας γιατί ήθελαν να χρηματοδοτήσουν ε, προγράμματα για τις σχέσεις ε, μεταξύ πόλεων και έπρεπε να τους απαντήσουμε ότι δεν υπήρχαν επαρκείς πόροι για να κάνουμε αυτά που επιθυμούσαμε. Οπότε η νέα πρόταση σε πρώτη άποψη από την πλευρά μας έχει βεβαίως φως αλλά και πολλές σκιές. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω το λόγο απευθείας στην κυρία Σιγκάν για να μας παρουσιάσει ακριβώς ποια είναι τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης ε, αξιολόγησης και σε τι βαθμό τα αποτελέσματα αυτά έχουν ληφθεί υπόψη για το νέο πρόγραμμα εάν δηλαδή θα είναι δυνατόν να μου εξηγήσετε μήπως τα κατάλαβα όλα λάθος, ίσως, μέλλον, ίσως μάλλον στο μέλλον το πρόγραμμα αυτό να βελτιωθεί. Κυρία Σιγκάν, έχετε το λόγο. Δέκα λεπτά παρακαλώ, για να έχουμε και λίγο χρόνο για συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας ε, παρουσιάσω και να συζητήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά έγγραφα γιατί όντως τον Απρίλιο και Μάιο φέτος δημοσιεύθηκαν πολύ σημαντικά έγγραφα για τα θέματα αυτά. Καταρχήν τον Απρίλιο είχαμε την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και η έκθεση που προβλέπει ο κανονισμός ε, και θεσπίζει την Επιτροπή είναι κάτι που μας αποσχόλησε για πολύ καιρό, προετοιμαστήκαμε πολύ καλά και ένα από τα στοιχεία που μας βοήθησε στην προετοιμασία είναι το ψήφισμα το δικό σας, το ψήφισμα της Επιτροπής σας που εγκρίθηκε πέρυσι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης είχαμε και δημόσιες διαβουλεύσεις που κράτησαν ε, αρκετούς μήνες ε, και έτσι δόθηκε ευκαιρία στους πολίτες να σχολιάσουν αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε πέρυσι και επεκτάθηκε σε φέτος το πρώτο εξάμεινο. Επίσης είχαμε και μια εξωτερική αξιολόγηση και εμείς σε επαφή με τα εθνικά σημεία επαφή και με τους ε, ενδιαφερομένους ε, εκπονήσαμε και τη δική μας αξιολόγηση που προσαρτήθηκε, επισυνάφθηκε μάλλον στην ανακοίνωση. Οπότε οι αξιολόγηση ήταν πολύ εμπεριστατωμένοι. Τον Απρίλιο υπευλήθη το σχετικό έγγραφο ε, ως προς την ουσία της δράσης και του στόχους του προγράμματος αλλά και ως προς τα ειδικά χαρακτηριστικά του επιβεβαιώθηκε με το παραπάνω ότι ε, γενικώ παίζει πολύ θετικό ρόλο το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των πολιτών και την δημοκρατική τους ε, ε, αν συμμετοχή και ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν ε, στην Ευρώπη και βοηθά στην ε, προώθηση της ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής και μακροπρόθεσμα και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα αυτό πρωτοπαρουσιάστηκε το 2012 για να αντιμετωπιστεί η κρίση εμπιστοσύνης και η περιορισμένη εμπιστοσύνη επιφυλακτικότητα προς τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, προωθώντας το μεγαλύτερο αίσθημα του ανήκειν ε, του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρουσιάζοντας τα πλεονεκτήματα της ε, ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα συμβάλλει ε, στην καλύτερη κατανόηση της ιστορίας, της πολυμορφίας, της πολιτιστικής διαφορετικότητας και βελτιώνει τις συνθήκες για συμμετοχή, δημοκρατική συμμετοχή του πολίτη. Εξακολουθεί να έχει αξία το πρόγραμμα και σήμερα, γιατί είχε σχεδιαστεί πριν από πολλά χρόνια για συγκεκριμένο σκοπό, αλλά εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό εργαλείο και έχουμε πει επανειλημμένως ότι το πρόγραμμα αυτό έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα, έχει επιμέρους προγράμματα για το ολοκαύτωμα, τη μνήμη του ολοκαυτώματος, επίσης ε, συνεργασία όσο ό,τι αφορά την αδελφοποίηση πόλεων. Όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία καθιστούν ιδιαίτερα ε, μοναδικό αυτό το πρόγραμμα. Κάτι που έδειξε η διάμεση αξιολόγηση είναι πόσο θετικό είναι το πρόγραμμα αυτό και ως προς την ουσία του και ως προς το γεγονός ότι επιτελεί το στόχο του το στόχο για τον οποίο σχεδιάστηκε. Ένα επιπλέον στοιχείο και θετικό για τα χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι ότι σε σχέση με άλλα προγράμματα χρηματοδότησης που αφορούν άμεσα πολιτικέ ευρωπαϊκή ένωση, το συγκεκριμένο πρόγραμμα καλύπτει ένα κενό, γιατί εξυπηρετεί τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ε, στοχεύει απευθείας προς τους πολίτες και αποτελεί ένα μοναδικό φόρουμ επαφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Ευρωπαίους πολίτες. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα του προβλήματος. Ήταν πολύ θετικό το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Με βάση τους δείκτες ε, όμως που χρησιμοποιήθηκαν από τον αρχικό κανονισμό, να σας δώσω κάποια σύντομα στατιστικά στοιχεία σε ό,τι αφορά την περίοδο 2014-2016 μια ναι, και πρόκειται για διάμεση αξιολόγηση. Πάνω από 7.000 σχέδια ε, ζητηθήκαν και έλαβαν χρηματοδότηση ή μάλλον υπευλήθησαν αιτήσει ε, για επιδοτήσεις. 7.000 σχέδια και πάνω από 1.000 σχέδια τελικά εγκρίθηκαν από 33 χώρες συμμετοχής. Σε ό,τι αφορά τους δείκτες που προτείνει ο κανονισμός, με τη χρήση αυτών των δικτών διαπιστώσαμε ότι ε, κάθε χρόνο αγγίζουμε ουσιαστικά με τα σχέδια αυτά πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες για αυτή την περίοδο 2014-2016. Και α, 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν άμεσα επηρεαστεί από το πρόγραμμα έμεσα μάλλον, 3 ε, εκατομμύρια άμεσα, 4 εκατομμύρια έμεσα. Βλέπετε, είναι τεράστια η απήχηση και η επιρροή του προγράμματος, ε, γιατί αγγίζει μεγάλο αριθμό πολιτών, άμεσα και έμεσα, με σχετικά χαμηλό κόστος. Γιατί ξέρουμε ε, τι σπάνιση υπάρχει πόρων. Αν έχουμε 7.000 αιτήσει για επιδότηση και έχουν εγκριθεί πάνω από 1.000 σχέδια, βλέπετε ότι παρόλα αυτά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε. Τώρα, τι κάνουμε με τη διαχείριση. Ε, σε συνεργασία με, την εκτελεστική, με τον εκτελεστικό οργανισμό προσπαθούμε να πλουστεύσουμε τις ε, διαδικασίες. Έχουμε προτείνει στο μεταξύ και τον πολιετή προγραμματισμό ώστε να εξασφαλίσουμε την απαραίτητη ελαστικότητα. Και σίγουρα το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες έχει αποδείξει την προστιθέμενη αξία του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχει στα μέλη του, στους συμμετέχοντες, αλλά και ως προς το συμπληρωματικό ρόλο που έχει σε σχέση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα και πολιτικές ε, ε, που αφορούν τον πολιτισμό, την παιδεία και την ιδιότητα του πολίτη. Τώρα, εντοπίσαμε και κάποιες άλλοι θα έλεγαν αδυναμίε, εμεί θα λέγαμε τομεί που επιδέχονται βελτιώσει. Κυρίω το πρόβλημα τη προβολή. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προβολή του προγράμματο, ώστε να γίνει πιο ορατό. Και επίση ε, θα πρέπει να εξετάσουμε ένα πιο φρέσκο πνεύμα αυτού του δείκτε. Να μην χρησιμοποιούμε σωρευτικά όλου του δείκτε, γιατί προτάθηκαν σε μια διαφορετική στιγμή. Και να δούμε τι συνέργειε υπάρχουν και τι συμπληρωματικότητα με άλλα προγράμματα που επίσης αφορούν ε, γενικώ την ηθαγένεια ή την έννοια του πολίτη. Και εδώ τώρα περνάω στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης που αφορά το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Δικαιοσύνη, τα Δικαιώματα και τις Αξίες. Γιατί όταν μιλήσαμε για προστιθέμενη αξία, ε, ξεκινήσαμε τις διαπραγματεύσεις με βάση κάποια αξιώματα. Το βασικό αξίωμα ήταν να βρούμε την προστιθέμενη αξία του προγράμματος για να δούμε πού θα το εντάξουμε στη νέα αρχιτεκτονική. Και επίσης ε, θέλησαμε να αποδείξουμε ότι προβάλλοντας το πρόγραμμα με τον τρόπο που το κάναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θέλησαμε να αποδείξουμε ότι οι προσπάθειές μας ανταποκρίνονται στην αναζήτηση συνεργειών και συμπληρωματικότητας και μιας προσπάθειας εξορθολογισμού ώστε να βρούμε κάποια κοινά σημεία και να διευκολύνουμε το σχεδιασμό και την όλη δομή του προγράμματος και να συμβάλλουμε και στην καλύτερη εκτέλεση, εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό ήταν ο πρωταρχικός στόχος ε, της προσπάθειάς μας, του εγχειρήματο αυτού. Και ένα από τα βασικά έγγραφα που χρησιμοποίησαμε για τη διαδικασία αυτή είναι ακριβώς η έκθεση για την ενδιάμεση αξιολόγηση που ήταν πολύ επίκαιρη και μια και ήταν το αποτέλεσμα πολύ σημαντικών συρρισφορών από πολλούς ενδιαφερόμενους και από τη δική σας επιτροπή. Είχαμε πολύ ε, βάσιμα επιχειρήματα για την όλη συζήτηση. Πάντως μπορούμε να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για το πρόγραμμα αυτό ε, που αφορά διάφορες δραστηριότητες ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά δικαιώματα αξίες, προωθεί ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί συμβάλλει στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και συμμετέχει στην ανάπτυξη μιας συμμετοχικής δημοκρατίας και μεγαλύτερη συμμετοχή στο Ευρωπαίο πολίτη, κάτι που είναι το ζητούμενο. Αποτέλεσμα του εγχειρήματο ήταν ότι συνδυάσαμε τα δύο προγράμματα, ε, το δικό μας για τα δικαιώματα και τις αξίες και το δικαίωμα της, ε, DigiJust για την ισότητα των δικαιωμάτων. Και τα δύο προγράμματα έχουν, ε, στο, έχουν στόχο τον Ευρωπαίο πολίτη, την κοινωνία των πολιτών και φυσικά θα εξαρτηθεί και από την εφαρμογή, αλλά θέλουν, επιδιώκουν τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Και σίγουρα η Επιτροπή σας τάχθηκε υπέρ του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες τα τελευταία χρόνια και τα επιχειρήματά που τα λάβαμε υπόψη και στη συζήτηση για την εφαρμογή του προγράμματος, την προετοιμασία του ψηφίσματος, αλλά και στη συνέχεια όλα αυτά τα όλη αυτή η συνεισφορά της Επιτροπής σας ήταν πολύ χρήσιμη για την αξιολόγηση που πραγματοποίησαμε. Μας ε, βοηθήσατε πολύ. Και μπορώ να πω ότι στην πρόταση ο σχεδιασμός του προγράμματος είναι τέτοιος όπου οι δράσεις του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες θα ακολουθήσουν την παρακαταθήκη και θα αξιοποιήσω την παρακαταθήκη του προηγούμενου προγράμματος η Ευρώπη για τους πολίτες. Και όλες οι δράσεις που έχουν ξεκινήσει, οι οριζόντιες δράσεις και η μεθοδολογία του νέου προγράμματος ε, είναι η φυσική συνέχεια του προηγούμενου. Ε, προτείνουμε συμμετοχή και ανάμειξη των πολιτών με δύο προτεραιότητες που ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τους στόχους του παρόντος προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες, κάτι που θα εξασφαλίσει μια φυσική συνέχεια των ε, δράσεων μετά την διάμεση αξιολόγηση του τρέχοντος προγράμματος. Σε κάποιο βαθμό μπορούμε να πούμε, βέβαια θα εξαρτηθεί όπως είπα και από την εφαρμογή, μπορούμε να πούμε λοιπόν σε μεγάλο βαθμό ότι οι νέοι άξονες θα προσφέρουν στο πρόγραμμά μας για τους πολίτες ε, ε, τη δυνατότητα να αυξήσουμε το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθεί και να, να διαφυλάσει τις αξίες, χρησιμοποιώντας την πράξη και τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα. Γιατί οι προτάσεις μας ε, φυσικά εδράζονται και στην αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος. Ε, και οι συνάδελφοι που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, συμμετείχαν στη συζήτηση και αυτό που κάναμε στη θεωρία πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί και εμπράκτος. Αυτό που ισχύει και για, το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες είναι ένα πρόγραμμα άιθαλες, ε, έχει διαχρονική αξία, είναι πάντα της μόδας και πάντοτε χρήσιμο και επίσης ε, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και μέλλοντος. Και πιστεύουμε ότι με την εφαρμογή του προγράμματος θα αγγίξουμε τη νεολαία. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία μας, όπως φαίνεται και από την ενδιάμεση αξιολόγηση. Και τώρα, να αναφερθώ σε τέσσερις ε, παρατηρήσεις ε, που ανταποκρίνονται σε δικά σας ε, αιτήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το πρώτο αφορά τον πρωταγωνιστικό ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες θα ενισχύσει τις δυνατότητες και τη χρηματοδοτική ε, αρρωγή προς την κοινωνία των πολιτών, δίνοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στη σε μη κυβερνητικέ οργανώσει ό,τι αφορά την προώθηση, τη διαφύλαξη και την ευαισθητοποίηση για τι ευρωπαϊκέ αξίε. Και συμβάλλει στο να μπορεί ο πολίτη να απολαύσει πραγματικά τα δικαιώματά του. Και ευθυγραμμίζεται πλήρω με τους στόχους του στόχου του ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του, τρέχοντος, του Απριλίου του τρέχοντο έτου. Γιατί σίγουρα προωθούν και υπερασπίζουν αυτέ τι αξίε οι ΜΚΟ. Ε, είμαι ιδιαίτερη περήφανη για τις συζητήσεις που είχαμε για το θέμα αυτό, το δεύτερο ζήτημα, τη νομική βάση που συζητήσαμε επανειλημμένως και δεν ήταν καθόλου εύκολο θέμα, γιατί προσπαθήσαμε με τα στοιχεία που προτείναμε στο σχεδιασμό του προγράμματος να δούμε πώς θα τα συνδυάσουμε με, τις, ε, με τη νομική βάση των συνθήκων. Στην προηγούμενη μορφή του το πρόγραμμα δεν καθιστούσε δυνατό κάτι τέτοιο δεν μπορέσαμε να συμπληρώσουμε τη νομική βάση με τον τρόπο που επιδιώκαμε όλοι. Αλλά τώρα στο νέο πρόγραμμα μπορέσαμε να βρούμε κάποιες διατυπώσεις και στο βασικό κανονισμό και στο παράρτημα που περιγράφουμε τις δράσεις, ώστε να συνδυάσουμε πολλές νομικές βάσεις. Πάντως το γενικό αποτέλεσμα μας δίνει μια νομική βάση που αντιμετωπίζει ισότιμα του δύο βραχίων στο νόμο παρασκευαστικού έργου, δηλαδή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Σύμβουλιο. Τώρα, το οικονομικό θέμα, πολύ σημαντικό, το αναφέρατε κι εσείς. Εδώ θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε οποιαδήποτε περικοπή των κονδυλίων. Το Ταμείο για τα Δικαιώματα και τις Αξίες προτείνει 947 εκατομμύρια για μία επτά αιτία 642 εκατομμύρια προβλέπονται για τα δικαιώματα και τις αξίες, το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και τις αξίες και 305 εκατομμύρια προτείνονται για το σκέλος δικαιοσύνη του προγράμματος. Επίσης είχαμε αύξηση κατά 16 εκατομμύρια για τα δικαιώματα και τις αξίες και μικρή αύξηση για τη δικαιοσύνη, ενώ η πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προβλέπει 233 ε, για τη συμμετοχή των πολιτών Κάτι δηλαδή που συνιστά μια μικρή δημοσιονομική αύξηση, όπως είπατε κι εσείς. Τώρα, να λάβουμε ως σημείο αφετηρίας, ως αναφορά μάλλον στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το βασικό επιχείρημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις διαπραγματεύσεις, σίγουρα ε, υστερούμε σε σχέση με τις προσδοκίες μας. Πάντως, ε, ως αφετηρή είναι πολύ καλή πρόταση, γιατί υπάρχει μια μικρή αύξηση και όλα φυσικά θα εξαρτηθούν από την πορεία των διαπραγματεύσεων και τη εξέλιξη της συζήτησης για την εφαρμογή του προγράμματος. Και θα δούμε πόσο θα προβληθεί το πρόγραμμα σε αυτή την πολύ σημαντική περίοδο. Γι' αυτό έχω ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε αυτή τη φάση του έργου για το νέο πρόγραμμα. Εφόσον η ενδιάμεση αναθεώρηση ασχολείται με κάποιου τομεί προ βελτίωση. Φροντίζουμε στο νέο πρόγραμμα να τα λάβουμε υπόψη μα. Γιατί οι δράσει, οι δραστηριότητε και ο τρόπο που διαμορφώνεται η συνεργασία μα ε, δεν έχει περάσει στην νομοθετική πράξη ακόμα σε αυτή τη φάση. Θα περάσει όμω από εσά και την εξέτασή σα και λαμβάνουμε υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν την προβολή, του δείκτε και άλλα στοιχεία που προανέφερα. Θα τα βρείτε και στην ανακοίνωση και αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως στοιχεία για τη βελτίωση και τη συνέχεια. Ε, και τώρα, ξεκινώντας σήμερα μαζί σας, ε, θέλουμε να παρουσιάσουμε το σχέδιο πρότασης που βρίσκεται επιτάπητος σε σχέση με την ενδιάμεση αναθεώρηση που και αυτή το αξίζει στους ε, ψηφοφόρους μας. Αύριο θα έχουμε διάλογο με τους πολίτες, με ενδιαφερομένους δηλαδή, βάσει του ισχύοντος κανονισμού. Ετησίως προβλέπεται αυτό και αύριο είναι ο επόμενος γύρος. Θα μιλήσουμε για το παρελθόν και για το μέλλον. Και με συγκεκριμένα στοιχεία όπως την, την προπαρασκευή της όλης διαδικασίας στο Κοινοβούλιο, εκδηλώσεις στον χώρο των πολιτών. Πολλά προβλέπονται ήδη και ένα τμήμα θα αφορά το να συζητήσουμε τα στοιχεία για τους τρόπους εφαρμογής του πρόγραμματος από τεχνική σκοπιάς, δηλαδή feedback ε, και αντιδράσεις προς τους από τους δικαιούχους για την απλούστευση και την ε, ε, χορήγηση των δωρεών και των δράσεων. Τέλος, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, βαδίζοντας τα τελευταία βήματα αυτής της διαδικασίας και όπως είπατε πρόεδρε θα εξαρτηθούν όλα από την εφαρμογή. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να είμαστε προσεκτικοί για να μην χάσουμε καμία φάση της διαδικασίας. Για να πετύχουμε όσα έχουμε ήδη επιτύχει μια φορά και με ακόμη περισσότερες δυνατότητες για βελτίωση. Σας ευχαριστώ, ελπίζω ότι έμεινα στα 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι η αξιολόγηση δείχνει ότι το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα επιτυχημένο, αλλά το ποσοστό εγκρίσεων που είναι λιγότερο από 10% δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Ως Κοινοβούλιο, με το ψήφισμά μας το Μάρτι, λοιπόν, είχαμε δίκιο, λέγοντας ότι θα θέλαμε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια ούτως ώστε αυτό το παιδί να γίνει επιτυχημένο. Και το πρόβλημα επίσης είναι, που μας δυσχεραίνει, είναι ότι διευρύνεται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής σε σχέση με το προηγούμενο, άρα η αύξηση είναι ακόμη πιο σχετική. Οπότε αυτό που μας παρουσιάζεται ως αύξηση ε, θεωρώ ότι δεν πολύ ισχύει, αλλά θα δούμε. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, θα ήθελα να πω να υποδεχθώ 14 ε, εκπαιδευόμενους από την ε, Γενική Διεύθυνση ΕΡΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ελπίζω η συζήτηση να σας προκαλεί ενδιαφέρον. Λοιπόν, να δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτριά μα την κυρία Σιλβί Γκυγιόμ. Εμείς εδώ έχουμε τη διαδικασία ping-pong. Μετά την Σιλβί Γκυγιόμ θα μπορέσετε εσείς να απαντήσετε. Και κατόπιν θα είναι συνάδελφο ε, Γιουνέ Μπαμπά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου. Σας ευχαριστώ κυρία Σιγκάν για την παρουσίασή σας. Ναι, πολλές ιδέες έχουμε όλοι και θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα με αυτό το πρόγραμμα για την Ευρώπη των πολιτών. Είναι πραγματική προστιθέμενη αξία με την ευρία έννοια. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Μιλήσατε για την ορατότητα του νέου προγράμματος. Απόλυτα θεμελιώδες αυτό. Αλλά ποια είναι η γνώμη μου. Νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να αποδυναμωθεί ε, το πρόγραμμα έτσι όπως το παρουσιάζεται. Πολλά λέγονται. Αλλά δεν βλέπουμε δηλαδή τι έννοια έχει αυτός ο συνδυασμός διαφόρων στοιχείων. Το αποκαλέσατε εξορθολογισμό των προγραμμάτων. Αλλά μήπως τελικά αυτό ήταν το κύριο στοιχείο για το καθορισμό του προγράμματος και όχι η λογική. Να σα δώσω ένα παράδειγμα. Λέτε ότι το θέμα τη ηθαγένεια δεν υπάρχει πλέον στον τίτλο. Ακόμη και συμβολικά έχει σημασία αυτό. Αυτό βοηθάει την ορατότητα προς τα έξω ή την ξυρίζει. Σαν τσουγκράνα. Είπατε ότι ήταν περίπλοκη η νομική βάση. Η επίτευξη της νομικής βάσης. Αλλά εγώ νομίζω πως ε, είναι καλό αυτό που επιτύχαμε. Το ότι θα συμμετέχει δηλαδή πλήρως το Κοινοβούλιο στην νομοθετική διαδικασία. Τώρα κάποιες ερωτήσεις. Τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Θα επιχειρήσω να είμαι σύντομη. να ξεκινήσουμε με τον προπολογισμό. Πρέπει να υπάρξουν κάποιε διευκρινήσει. Είπατε ότι προτείνετε το status quo. Το 2017 θα συμφωνεί και η Τερέζα νομίζω. Είχαμε ζητήσει μέσω ψηφίσματος ε, αύξηση της χρηματοδότησης. Δεν νομίζω ότι την έχουμε επιτύχει. Και επειδή υπάρχει πολλή απογοήτευση για το πρόγραμμα αυτό, δεν θα έπρεπε αυτή η απογοήτευση να αυξηθεί ακόμη περισσότερο. Ίσως θα πρέπει να έρθετε και στο θέμα της κατανομής. Πώς θα κατανεμηθούν τα ποσά μεταξύ των διαφόρων δράσεων. Θέλουμε διευκρινήσεις. Τώρα για να το πω λίγο χοντρικά. Τι εννοείται αξίες. Πώς θα τις παρουσιάσετε. Τώρα τα παρουσιάζω λιγάκι χοντρά. Τον ένα χρόνο θα προωθήσουμε την ε, ισότητα, τον επόμενο χρόνο την ε, πολυμορφία. Πώς θα συνδυαστούν και ποια είναι η, ε, η ταξινόμησή τους, πώς θέτουμε τις προτεραιότητες. Τρίτον, επικοινωνία. Θέλουμε να είναι πιο παρούσα η επικοινωνία, αξιοποιώντας και τα ψηφιακά μέσα. Τι εννοεί όμως το άρθρο 18 που λέει ενημέρωση και δημοσιεύσεις. Όλα αυτά περνάνε και μέσα από τη θεσμική ενημέρωση για τους στόχους της Ένωσης, λέτε. Αλλά θα στηρίξουμε έτσι τα τοπικά προγράμματα, δηλαδή τις ε, καμπάνιες, οι καμπάνιες ενημέρωση των θεσμών έχουν ήδη επαρκείς πόρους. Μήπως τα μπερδεύουμε. Χρειάζονται ευκρινήσεις. Και για το άρθρο 7. Λέτε ότι θα ανοίξουμε το πρόγραμμα και με προς τις συνδεδεμένες τρίτες χώρες. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα υπάρξει περαιτέρω διασπορά των πόρων. Πώς θα το εφαρμόσουμε αυτό. Ποιες άλλες χώρες. Η προσένταξη θα είναι. Ή ποιε. Και σε άλλα σημεία θέλω διευκρινήσει. Λέτε θα χρηματοδοτήσετε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και διάφορα άλλα προγράμματα των πολιτών. Τα είπαμε και πέρυσι. Θέλω να είμαστε πιο συγκεκριμένοι πώς θα στηρίξουμε και φορείς και τοπικές πρωτοβουλίες για να υπάρξει μια σωστή κατανομή μεταξύ αυτών. Ούτως ώστε η επιλογή, για παράδειγμα, ποιες μήκυο θα χρηματοδοτήσουμε, η επιλογή να γίνει με σαφή κριτήρια. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολλά άλλα για το Εθνικό Σημείο Επαφής και τα λοιπά. Ναι, τελειώνω. Και για το ρόλο που θα μπορούσε να έχει το Κοινοβούλιο για το καθορισμό των προτεραιοτήτων. Και κάτι ακόμη προς την πρόεδρό μας. Γενικά δεν μπαίνω σε θέματα σύγκρουση αρμοδιοτήτων άρθρα 54-55 είναι πολύ ολιστηρό αυτό το πεδίο αλλά θα παρακαλούσα την Πρόεδρο να επαγρυπνεί ούτω ώστε να έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για το σημείο Β. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σιλβί. Μα σε διαβεβαιώ ότι το έχουμε ήδη κάνει αυτό. Έχουμε αποκλειστική αρμοδιότητα για το τμήμα αυτό και το πρόγραμμα είναι σαφώς τόσο διαρθρωμένο ούτω ώστε οι διάφοροι τομείς του να είναι σωστά οριοθετημένοι. Και ελπίζω ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα με τη Λίμπε. Αλλά θα δούμε βέβαια. Κυρία Σιγκάν, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Γκυγιόμ. Βρισκόμαστε συχνά και στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Απλώ για το γεωγραφικό πεδίο που αναφέρατε και εσείς κυρία Πρόεδρε στην αρχή. Θα σας καλέσω να δείτε και θέλω να το πω και εξ αρχή. Μετά μπορούμε να οργανώσουμε και τεχνικές συνεδριάσεις. Για να μπούμε στις λεπτομέρειες αν θέλετε, τώρα δεν είναι δυνατόν. Ως προς την γεωγραφική κατανομή των προγραμμάτων στην δική αξιολόγηση υπάρχει ένα κεφάλαιο συγκεκριμένα για το τι έχει γίνει με τα προγράμματα ως τώρα, τη γεωγραφική τους κατανομή και σε όλες τις χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε έχουμε προγραμμα, προγράμματα. Απλώ η κατανομή δεν είναι πάντοτε ε, ισορροπημένη. Ε, υπάρχει περιγραφή του σχετικού θέματος. Αυτό για το γεωγραφικό πεδίο και για να ολοκληρώσω το πρόγραμμα τώρα ε, αρχίζει να εφαρμόζεται στα Αρκτικά Βαλκάνια. Και θέλουμε και να συνεχίσουμε. Αλλά αν τα συνδυάσουμε αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα και για το μέλλον σε περίπτωση που εφαρμόσουμε σε τρίτε χώρε. Προβολή. Για την προβολή, εάν κοιτάξετε το παράρτημα 1 της πρότασης, στο σημείο K, εδώ μπορούμε να ενισχύσουμε την γνώση περί του προγράμματος, τη διάδοση των αποτελεσμάτων του και την προσέγγιση των πολιτών με τα εθνικά δίκτυα επαφής. Αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Ε, ο μηχανισμός μας και η διαπλοκή μας με κράτη-μέλη, με ε, πολίτες και ενώσεις τους, με, τις, με τους κρατικούς φορείς, δηλαδή η συνεννόησή μας με όλους αυτούς, είναι τέτοιας μορφής που μπορείτε να το δείτε και με συγκεκριμένα παραδείγματα για το πώς επικοινωνούμε. Έχουμε κάνει βήματα για να ενισχύσουμε την προβολή στα σημεία εθνικής ε, τα εθνικά σημεία επαφή, με τη σχετική πλατφόρμα για την προβολή των αποτελεσμάτων του προγράμματο. Στην ενδιάμεση αξιολόγηση έχουμε συμπεριλάβει ε, τη σχετική διάσταση για την προβολή. Αξίες. Δεν υπάρχει ιεράρχηση των αξιών Και το καταλαβαίνω, είχαμε έναν ωραίο κανονισμούλι όπου όλα ήταν ε, πολύ σωστά διαρθρωμένα περί του προγράμματος και καταλήξαμε τώρα με το νέο σχέδιο. Εάν το διαβάσουμε, το μελετήσουμε και το καταλάβουμε καλύτερα, θα δούμε όλοι, γιατί συμμετείχαμε επί μακρόν, στις δυναμικές και εκβάθρων διαπραγματεύσεις για την κατάσταση του κανονισμού. Εάν λοιπόν τα κάνουμε όλα αυτά, θα καταλάβουμε ότι το κείμενο χρειαζόταν ευθυγράμμιση. Πρέπει να υπάρχει οικονομική εκπροσώπηση και η αλλαγή που έχει γίνει δεν είναι τόσο πολύ στην ουσία. Το αντίθετο. Σα διαβεβαιώ ότι όλε οι δραστηριότητε που καλύπτονται από το Ευρώπη για του πολίτε και όλοι οι τρόποι συνεργασία μα περιέχονται σε αυτό το κείμενο. Ίσως θα ήταν ευκολότερο να υπάρχουν όλα σε ένα συγκεκριμένο άρθρο, επειδή όμω ο σκοπό τη όλη αυτή τη προσπάθεια ήταν να είμαστε συνεπεί ευθυγραμμίζοντα και διαμορφώνοντα σχέσει συνεργασία ήταν αδύνατο να συνδυάσουμε δύο στοιχεία και να τα βάλουμε το ένα μετά το άλλο διαδοχικά. Η συζήτηση ήταν πιο περίπλοκη. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και μετά θα έχουμε και τεχνικότερες συναντήσεις κατά πόσον τα στοιχεία αυτά είναι πιο σκόπιμα για αυτό το βήμα συζήτησης παρά από την ίδια την ουσία του θέματος. Θα συνεχίσουμε όμως γιατί έχουμε δυνατότητες βελτίωσης. Για τον προπολογισμό. Όσα λέτε μου φαίνονται εξαιρετικά. Πάντοτε παρακολουθώ τις συστάσεις σας. Για τον προπολογισμό που εσείς θεωρείτε τον καταλληλότερο στο το πρόγραμμα να έχει ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα και μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γι' αυτό λοιπόν μόνο συνεργασία μπορώ να σας ε, υποσχεθώ για τα επόμενα βήματα κατάρτισης του προπλογισμού και για την, για την επικοινωνία νομίζω το ανέφερα. Για τα τοπικά προγράμματα, για την τοπική διάσταση όλου αυτού του θέματος. Στο σχέδιο αυτό καταφέραμε για τις ευρωπαϊκές πόλεις να συμπεριλάβουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Μας βοήθησε αυτό να διατηρήσουμε τα μενοδικά χαρακτηριστικά του προγράμματος που επιτρέπουν στα μικρά προγράμματα και έργα να περάσουν στο τοπικό επίπεδο, επιτόπου, για να είναι κοντά στους πολίτες. Αυτό το είπα από την αρχή. Η ουσία του προγράμματος, πιστεύω, διατηρείται και όλα αυτά τα στοιχεία που κάνουν αυτό το πρόγραμμα τόσο μοναδικό υπάρχουν στο σχέδιο του κειμένου. Θα αξιοποιήσουμε όμως το δυναμικό της νέας πρότασης, διότι υπάρχει αυτό. Απλώς πρέπει να το εντοπίσουμε και να το υλοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Τρία λεπτά σε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την κυρία Θήγκαν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ευρώπη για τους πολίτες και ευχαριστώ και το συντάκτη της μελέτης ε, που μας έστειλε το Τμήμα Πολιτικής Β την εβδομάδα αυτή για τα επιμέρους προγράμματα. Είμαι σκιώδης ηγετρία σε ένα πρόγραμμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα γιατί πιστεύω πραγματικά σε αυτό το πρόγραμμα Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα μιλήσαμε για σταθερή χρηματοδοτική αύξηση. Τελικά φαίνεται ότι με τη νομική βάση βρέθηκε η λύση από τα, από τα 185 εκατομμύρια να φτάσουμε στα 203. Καλή αύξηση, αλλά εμεί είχαμε ζητήσει 500 εκατομμύρια, οπότε είναι σχετικά μικρή σε σχέση με τις δικές μας προσδοκίες. Πώς θα συνδυάσουμε αυτό το πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, δικαιώματα και αξίες χωρίς να χάσουμε τμήμα της προσωπικότητας αυτού του προγράμματος, γιατί στην πορεία αυτό χάσω, χάσαμε, γιατί επρόκειται για ένα πρόγραμμα που μιλούσε άμεσα για τους πολίτες. Ήδη το, ο τίτλος του προγράμματος περιλάμβανε και τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα δεν αναφέρονται. Μήπως ε, χάσουμε κάτι από την ουσία του προγράμματος, ό,τι αφορά τα τοπικά σημεία επαφής και τους ε, υπεύθυνους. Ε, ε, αυτοί θα εκπροσωπήσουν και το ευρύτερο πρόγραμμα για τη δικαιοσύνη, τα δικαιώματα και, την και τις αξίες ή μόνο το σκέλος για την Ευρώπη των πολιτών. Νομίζω ότι ήταν λίγο απογοητευτικό αυτό. Αν και πιστεύω ότι το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να συνεχιστεί οπωσδήποτε και ελπίζω να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πόσο σημαντικά είναι τα θέματα που αφορούν τον πολίτη και πόσο σημαντικό έργο έχει επιτελεστεί μέχρι στιγμής. Σας ευχαριστούμε και καλή τύχη για την επόμενη φάση του προγράμματος. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Sigan. Sie haben das... Ευχαριστώ. Κυρία Σιγκάν, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Τι να πω, τι να πω. Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω το ίδιο μήνυμα. ό,τι υπάρχει στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες θα, θα διαφυλαχθεί. Και καταλαβαίνω τα σχόλιά σας, είναι αναμενόμενη η αντίδραση. Γιατί πρώτη πρώτης όψεως δεν βλέπουμε ε, την Ευρώπη για τους πολίτες. Πού είναι οι πολίτες. Θα πρέπει να ψάξουμε τη δομή για να τους αναζητήσουμε. Πάντως το καθήκον μας είναι, κυρίως το δικό μας είναι, αυτές οι διευκρινήσεις και η ενημέρωση να γίνει προς όλους τους ενδιαφερομένους, όλους που μέχρι τώρα είχαν κάποια σχέση με το πρόγραμμα, τους ε, ε τωρινούς αλλά και τους δυνητικούς δικαιούχους. Γιατί ενισχύουμε και νέες ε, του προγράμματος. Πάντως το παλιό πρόγραμμα διαφυλάσσεται πλήρως. Αναφέρθηκε και προηγουμένως στο παράρτημα 1 και το σημείο Κ και το πρόγραμμα για την στήριξη των εθνικών ε, σημείων επαφής. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα γιατί το σημείο αυτό έχει δοκιμαστεί και είναι πολύ χρήσιμο για την εφαρμογή του προγράμματος. Και όσο συνεχίζεται ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών, τόσο το καλύτερο. Και μάλιστα πολύ πιθανό να αυξήσουμε και τον αριθμό των συνεδριάσεων και επαφών κατά τη διάρκεια του έτους. Και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία με τα τοπικά σημεία επαφής. Και οι πιθανές συνέργειες θα εξαρτηθούν από το πώς οι διάφοροι τομείς καλύπτονται στα κράτη-μέλη. Γιατί αυτά ελέγχουν το διοικητικό σκέλος. Πάντως ό,τι μέχρι στιγμής έχει δοκιμαστεί και έχει αποδώσει καρπούς θα συνεχιστεί και στο νέο πρόγραμμα. Στην πρώτη φάση θα πρέπει να προωθήσουμε το μήνυμα ότι οι δράσεις ε, του προγράμματος ε, Ευρώπη και τους πολίτες ε, διαφυλάσσονται. Τώρα, αν το όνομα του προγράμματος είναι διαφορετικό στο μέλλον, ο τίτλος είναι κάπως διαφορετικός, αυτό είναι προσυζήτηση. Το πιο σημαντικό είναι να περάσει σε όλους το μήνυμα. Σε όλους, όχι μόνο στου είναι εξοικειωμένοι με το πρόγραμμα, αλλά και στους υπόλοιπους, ότι μπορεί το όνομα να έχει αλλάξει, αλλά οι δραστηριότητες παραμένουν και τα καλά σημεία θα διατηρηθούν, ενώ οι αδυναμίες θα διορθωθούν. Πρώτο λοιπόν μέλημά μας είναι να προωθήσουμε, να διαφημίσουμε κατά κάποιο τρόπο από κοινού το ισχύον πρόγραμμα με τις νέες του πτυχές. Ευχαριστώ κυρία Μπίλτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω επιφυλάξει όσον αφορά το πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες, γιατί έχει μια ιδεολογική χρειά. Για παράδειγμα, μνήμη. Η ευρωπαϊκή ιστορία αντιμετωπίζεται με απλουστευτικό τρόπο. Αντιμετωπίζει τον ολοκληρωτισμό, ε, αντιπαραθέτει τον ολοκληρωτισμό με μια ευρωπαϊκή ταυτότητα που είναι ανοιχτή στη μετανάστευση, ε, ενδιαφέρεται για την ε, πολιτισμικότητα. Δηλαδή, δεχόμαστε οτιδήποτε. <clears throat> Και οτιδήποτε δεχόμαστε τελικά καταλήγει στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Η κληρονομιά μας πρέπει να παρουσιάζεται θετικά. Να εμείνουμε στην συμμετοχή και τη συμβολή του χριστιανισμού. Τώρα για τις ε, δράσεις στον πολιτικό τομέα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να <clears throat> ε, ενισχύουμε ε, τις ομάδες που εργάζονται για τους, ε, για τους πιο ευάλωτους και ιδιαίτερα τους μετανάστες. Αυτό καταλαβαίνετε ότι μετά την Ουγγαρία και η Ιταλία μπορεί να νομοθετήσει για τις οργανώσεις για τη βοήθεια αυτές και πώς θα αντιμετωπίσετε τις, τους δισταγμούς των κρατών μελών για διάφορους φορείς γιατί θεωρείτε ότι παρεμβαίνουν ε, στην πολιτική, στα εσωτερικά των χωρών αυτών. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις παρεμβάσεις. Η κυρία Σιγκάν. Παρακαλώ διαβάστε την ενδιάμεση αξιολόγηση. Και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε τα διάφορα σημεία που περιέχει όπου συζητάμε και τα διμερεί και τα οριζόντια προγράμματα και τους στόχους του προγράμματος και τα αποτελέσματα εφαρμογής του προγράμματος τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά τα λέει αυτή η έκθεση. Να τα δούμε σημείο-σημείο για τα διάφορα στοιχεία. Γιατί δείχνουν και είναι αποτέλεσμα πολύ ευρείας αξιολόγησης δείχνουν ότι το πρόγραμμα όντω προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία σε όλους αυτούς τους τομείς. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να εξετάσετε αυτό το κείμενο για να δείτε μαζί μας όλα αυτά τα στοιχεία. Το πρόγραμμα θεωρείται πολύ καλό με βάση αυτήν την αξιολόγηση. Προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλη προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό θέλουμε να το συνεχίσουμε και γι' αυτό συμπεριλήφθηκε το πρόγραμμα αυτό και στο σχεδιασμό του προγράμματος για τις αξίες. Αλλά να τα δούμε ένα-ένα τα σημεία βεβαίως. Γιατί μελετώντας αυτή την αξιολόγηση των διαφόρων προγραμμάτων Εντάξει, εσείς κάνετε την ε, αξιολόγηση τη δική σας. Ίσως συμμετείχατε στη δημόσια διαβούλευση που είχαμε πέρυσι. Να τα εξετάσουμε μαζί τα έγγραφα αυτά, να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα. Και από το 2017 έχουμε μια πολύ ωραία συλλογή αυτών των προγραμμάτων. Αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος για να επιχειρήσουμε να σας πείσουμε για αυτό για το οποίο εμείς είμαστε ιδιαίτερα πεπισμένοι, ότι προσθέτει ιδιαίτερη αξία, που είναι ιδιαίτερα ευρεία. Ευχαριστώ πολύ. Σίλβια, δύο λεπτά. Απλώς να πω ότι η ομάδα μας αποδίδει άκρα σημασία στο πρόγραμμα αυτό. Είναι σημαντικό για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ε, απομάκρυνσης από την Ευρώπη, της υποβάθμισης της συμμετοχής των πολιτών, της αφοσίωσης της ε, ε, δράσης της κοινωνίας των πολιτών Βεβαίω συμφωνώ με πάρα πολλά από αυτά που είπε η Σιλβί Γκυγιόμ. Ήθελα απλώ να επαναλάβω τρία πράγματα. Ε, το πρώτο, ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και σωστή διαχείριση των δύο προγραμμάτων ε, που θα συνενωθούν και να μην υπάρξει σύγχυση στους ε, δικαιούχου που είναι συνηθισμένοι σε διαφορετικέ πηγέ από τις οποίες ενισχύονται. Υπάρχουν σημεία σύγκληση των προγραμμάτων, αλλά καλό είναι να υπάρχει μια καλή ε, γνώση των δύο προγραμμάτων χωρίς να υπάρξει σύγχυση όπως τώρα συμβαίνει για τον προπολογισμό τώρα. Ε, εμείς ως Κοινοβούλιο και Επιτροπή Πολιτισμού ε, είδαμε τα ανησυχητικά δεδομένα του προπολογισμού και είδαμε ότι στα προγράμματα της κοινωνίας των πολιτών υπήρξε 6% μόνον ε, πρόσληψη. Πολύ απογοητευτικό. Το πρόγραμμα αυτό είναι αυξανόμενο ενδιαφέροντος ωστόσο για τους πολίτες και Τρίτον, ήθελα να ξέρω τι γίνεται με το Valor Platform, την πλατφόρμα που θα γίνει ένα σημαντικό εργαλείο εργασίας ε, και μέθοδος για την διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Τι επενδύσεις γίνονται από αυτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Σιγκάλη. Πολύ μου άρεσε η έκφρασή σας με το management. Σωστό, αλλά είναι και φυσιολογικό το σχέδιο που αναζητά σχέσεις συνεργασίας, συνοχή, ευθυγράμμιση κλπ. Αυτά έχει. Αλλά εμείς ξέρουμε το δικό μας πρόγραμμα. Και την Ευρώπη για τους πολίτες εδώ. Είναι ένα θέμα λοιπόν για μα, αλλά τα γνωρίζουμε όλα αυτά τα στοιχεία, διότι τα διαπραγματευτήκαμε όλα. Εμεί φροντίσαμε να συμπεριλαμβάνονται σε πρώτη φάση. Ήταν όμω σαφέ και, από τι συζητήσει και ήταν και αναμενόμενο με ένα απλούστερο καινούριο έγγραφο να πρέπει να μπορούμε να εξηγήσουμε στο δημόσιο τομέα που είναι τα νέα στοιχεία του προγραμματός μας. Ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε τα νέα στοιχεία του προγράμματος για να προωθήσουμε ακριβώς το πρόγραμμα. Αυτό είναι το στοιχείο της ενημέρωσης από την άλλη και το στι... η διάσταση της υλοποίησης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε το πρόγραμμα ακόμα καλύτερα κιόλα. Συμφωνώ όμως απολύτως. Επίσης το θέμα της ε, μεικτής νομικής βάσης δεν ε, απλουστεύει τα πράγματα. Νομικός όμως ομιλώντας, ο μόνος τρόπος να συνδυαστούν τα στοιχεία στο σχέδιο με την σωστή νομική βάση ήταν αυτός. πρέπει να εξηγήσουν, να ε, συνδυάσουν τις δυναμικές βάσεις. Κάτι που ένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να το καταλάβει, από νομοθετικής άποψης είναι απαραίτητο. Έτσι έχει μια διαδικασία αναθεώρησης και έτσι είναι και η δημοκρατική προσέγγιση για αυτό το πρόγραμμα, για τον προπολογισμό. Δεν θα σχολιάσω ε, άλλο. Νομίζω τα στερέψανε τα σχόλια μου. Και για την πλατφόρμα, στην ενδιάμεση να σε ένα από τα κεφάλαια υπάρχει πληροφόρηση για τις λεπτομέρειες της πλατφόρμας αυτής και τα αποτελέσματα. Είναι κάτι σαν ε, online βάση δεδομένων για την ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή βελτιστών πρακτικών μεταξύ των δικαιούχων, των ε, πολιτών και των όσων συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό. Ε, Βοηθά λίγο στην υλοποίηση της λογικής της όλης ε, αναθεώρησης του προγράμματος. Θα μπορούσαμε να το παρουσιάσουμε λεπτομερέστερα και να το επεξεργαστούμε και περισσότερο. Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποιοι τομείς βελτίωση της ενδιάμεσης αναθεώρησης και εκεί φροντίζουμε να παρουσιάσουμε τα σχετικά προγράμματα με τα αποτελέσματά τους. Εδώ χρειαζόμαστε feedback και ανταπόκριση, απαντήσει από το κοινό, για να πιστούν για το ποια είναι τα ωφέλη του προγράμματο. Το ταξίδι λοιπόν, Το ταξίδι αυτό ελπίζουμε να πάει καλά και με τη δική σας βοήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα έχουμε ακόμη πολλές συζητήσεις τους επόμενους μήνες έχετε ένα συνδυασμό νομικών βάσεων. Χρειάστηκε να καταλήξετε σε κάτι τέτοιο. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι και άλλες επιτροπές θα θέλουν τώρα να έχουν δικαίωμα συναρμοδιότητας. Πρέπει να το λύσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Όμως σημαίνει ότι το σφιχτό χρονοδιόγραμμα που έχουμε μέχρι τέλους της κοινοβουλευτικής θητείας θα γίνει ακόμη πιο σφιχτό. Αλλά ελπίζω να βρούμε μια καλή λύση. Υπάρχουν πολλά θέματα λεπτομεριών που θα πρέπει να συζητηθούν μεταξύ των σκιωδών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τονίζω ότι σημαντικό είναι να υπάρχουν επαρκείς πόροι. Αλλά θα το συνδυάσω και με το ποσοστό απόρριψης. Γιατί αυτό δημιουργεί απογοήτευση στους ετούμενους. Ε, υποβάλλουν καλά προγράμματα και απορρίπτονται που είναι πολύ καλά και θα μπορούσαν να προωθηθούν, να εγκριθούν, αλλά δεν εγκρίνονται γιατί δεν υπάρχει πλέον ε, χρηματοδότηση. Αυτό αυξάνει την απογοήτευση, γιατί τα κράτη-μέλη δεν είναι δεδεθειμένα να πρικοδοτήσουν επαρκώς το πρόγραμμα, αλλά τελικά η απογοήτευση και η οργή στρέφεται κατά της Ένωσης. Μα αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει να επιτύχει το πρόγραμμα αυτό. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε από κοινού, ούτω ώστε τα προγράμματα αυτά να λάβουν περισσότερη χρηματοδότηση για να επιτύχουν τους στόχους. Γιατί αλλιώ οι απορρίψει επιτυχάνουν το αντίθετο. Θα ήταν απόλυτα λανθασμένο κάτι τέτοιο. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ για την παρουσία σα. Σίγουρα δεν είναι η τελευταία φορά. Θα επιχειρήσουμε λοιπόν από κοινού να το βελτιώσουμε αυτό το πρόγραμμα όσο γίνεται, ούτω ώστε να έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Και ελπίζω ότι θα αγωνιστείτε κι εσείς μαζί μας για να λάβει και επαρκή πρικοδότηση γιατί το πρόβλημα νομίζω ότι κυρίως είναι το Συμβούλιο. Ναι, τελικά θα δούμε τι θα γίνει, αλλά έχουμε πολύ σκληρή δουλειά μπροστά μας και συνολικά βέβαια για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλό απόγευμα. Θα τα ξαναπούμε. Οπότε, τελευταίο σημείο της μέρης της διάταξης που θα λάβει χώρα και κλεισμένο το θεό. Όσοι λοιπόν δεν είναι βουλευτές ή συνεργάτες του Κοινοβουλίου να αποχωρήσουν.